Καλημέρα σε όλους. Έχουμε εδώ όλες τις πολιτικές ομάδες έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Αντίθετα με τα όσα υπήρχαν στη ημερήσια διάταξή μας, η κυρία Ρουαπίζα η οποία είναι ε, αναπληρωτής ε, Γενική Διευθύντρια του του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου δεν θα μπορέσει να έρθει, οπότε θα την έχουμε μαζί μας σε μια επόμενη συνεδρίαση. Έχουμε τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης. Υπάρχουν κάποια σχόλια? Αν όχι, θεωρείτε ότι εγκρίνονται. Ανακοινώσεις, σημείο 3. Συνήθως, όπως συνήθως ε, θα μεταδίδεται στο ίντερνετ αυτή η συνεδρίαση. Έχουμε ήδη διανύμει τον αντίστοιχο κατάλογο. Θα καταλωσορίσω τώρα τον κύριο Φέλιξ Ρούτς, ο οποίος βρίσκεται στα δεξιά μου από την ε, Επιτροπή της Γραμματείας ε, και αντικαθαστεί τον Ανδρέ Κοράντο που ήταν μαζί μας ε, για τρία χρόνια. Αυτό είναι λόγω της, ε, των απαιτήσεων για κινητικότητα των υπαλλήλων στο Κοινοβούλιο. Καλώς ήλθατε στο κλαμπ. Πολύ απαιτητική η θέση που σας ε, δώσανε. Η Πορτογαλική τηλεόραση μου ζήτησε να τους δώσω κάποια κομμάτια της συνεδρίασής μας το απόγευμα. Έχετε κάποια αντίρρηση? Ο συνήθως δεν υπάρχει αντίρρηση. Σημείο 4. Ο κανονισμός για την πρόσβαση στην αγορά βγαίνει μια σειρά από χώρες ΑΚΕ από την, από κατάλογο των χωρών που έχουν καταλήξει σε διαπραγματεύσεις, στις διαπραγματεύσεις που σχετίζονται με τις, οικονομι... τις ε, συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης. Η θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια στις 17 Ιανουαρίου Άρα μπαίνουμε στην τακτική διαδικασία για τη δεύτερη ανάγνωση. Έχουμε ε, τρεις ε, μήνες εργασίας με μια πιθανή επέκταση για ένα μήνα. Θα εξετάσουμε τη θέση το Συμβουλίο, θα δούμε ποια είναι τα βήματα που θα ακολουθήσει το ε, Κοινοβούλιο. Ο Ντέβιτ Μάρτιν, ο εισηγητής, ε, δεν μπόρεσε να είναι εδώ γιατί θα πάει στην Ιορδανία με την Επιτροπή που παρατηρητών για τις εκλογές. Σήμερα είναι οι εκλογές και θα τον αντικαθαστήσει ο Ζορ Κούτας, στον οποίο δίνω το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους του Ντέιβιτ που δεν βρίσκεται σήμερα μαζί μας. Αλλά είμαι σίγουρος ότι θα παρακολουθήσει τα όσα θα υποθούν σήμερα στη συζήτηση. Να σας παρουσιάσω τώρα τα σχόλιά του. Μια σύντομη παρουσίαση της έκθεσης για να σας ε, θυμίσω. Ο κανονισμός για την πρόσβαση στην αγορά παρέχει ε, μία ε, προσωρινή πρόσβαση στη, για τις, ε, τους δασμούς στις χώρες που έχουν καταλήξει συμφωνία μέχρι το τέλος του 2007. Ο κανονισμός θεωρήθηκε μια προσωρινή λύση πριν από την κύρωση των ε, συμφωνιών για να αποφευχθεί κάποια διατάραξη του εμπορίου. Πρόκειται για μια πρόταση τροποποίησης κανονισμού της Κομισιόν ε, για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την εφαρμογή των συμφωνιών μέχρι τον Ιανουάριο του 2014. Το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του στην πρώτη ανάγνωση. Το Σεπτέμβριο του 2012 εγκρίθηκε στην Ολομέλεια. Τα βασικά ζητήματα ήταν μια τροπολογία για αναβολή της έναρξης ισχύω του κανονισμού αντί για 1η Ιανουαρίου του 2014 να πάει το 2016. Επίσης υπήρχαν τρεις ε, τροπολογίες για τις ε, πράξεις εξουσιοδότηση που εγκρίθηκαν στην ε, προπαρασκευαστική συνάντηση μιλήσαμε για την ανάθεση των εξουσιών και φαίνεται ότι αυτό σχετίζεται με τα όσα υιοθετήσαμε στο Omnibus 2. Το 2010, όπως είπε και ο Πρόεδρος, υπήρξε μια πολιτική συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση, η οποία εγκρίθηκε στις 11 Δεκεμβρίου του 2012 και ανακοινώθηκε στην τελευταία Ολομέλεια. Έτσι λοιπόν το Συμβούλιο υποστήριξε τις θέσεις ε, του Κοινοβουλίου μόνο με κάποια τεχνική προσαρμογή για τη Ζιμπάμπουε στο ε, πρώτο παράρτημα χώρες ε, που επωφελούνται γιατί μπήκε στην συμφωνία αφού έκανε την πρότασή της η Κομισιόν. Ήδη η συμφωνία με τη Ζιμπάμπου εμφαρμόζεται από το Μάιο και η αλλαγή από το Συμβούλιο ακολουθεί τη λογική του κανονισμού και της πρότασης της Κομισιόν. Το Συμβούλιο δεν υποστηρίζει καμία από τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου, ούτε και η Κομισιόν. Παρ' όλα αυτά σημειώνεται ότι η γαλλική αντιπροσωπεία είχε διαφορετική άποψη από τη δική μας. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε μια θέση στη δεύτερη ανάγνωση, τρεις, το ανώτερο τέσσερις μήνες στα διαρκέσει διαδικασία. Ο εισηγητής θεωρεί ότι θα ήταν χειρότερο να προσπαθήσουμε να βρούμε συμφωνία με το Συμβούλιο εκ των Προτέρων και γι' αυτό θα ήθελε να ζητήσει εντολή για να μπει σε άτυπες συζητήσεις με το Συμβούλιο και την Κομισιόν για αυτό το θέμα. Με βάση την εντολή, η βάση της εντολής θα είναι η θέση που εγκρίθηκε το Σεπτέμβρη πέρυσι, στην πρώτη ανάγνωση. Για να δούμε τώρα τι θέλουν να πούνε οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ. Τίποτα. Υπάρχει κάποιος που θα ήθελε να κάνει κάποιο σχόλιο για αυτό το θέμα. ο Σκιώδης. Την τελευταία. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος να επαναληφθεί η συζήτηση την οποία είχαμε στο παρελθόν γύρω από το θέμα αυτό. Το ερώτημα που τίθεται είναι τι θα πει προσωρινό. Πόσο κρατάει το προσωρινό. Μερικές φορές το προσωρινό διαρκεί πολύ περισσότερο από το μόνιμο. Νομίζω λοιπόν ότι εμείς θα υποστηρίξουμε σαν Ευρωπαϊκό Κόμμα την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν μας ε, δημιουργεί πρόβλημα η θέση του Συμβουλίου. Υπήρξε μια αρκετά μεγάλη μειονότητα, μειοψηφία συγγνώμη, στην Ολομέλεια που στήριξε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το θέμα που τίθεται είναι το πώς εμείς θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα εμείς πιστεύω ότι σε αυτή τη φάση δεν έχουμε την πολυτέλεια της καθυστέρησης. Μπορεί κανείς να διαπραγματεύεται για πάντα και ας ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις, αλλά το θέμα είναι ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση η διαφορά είναι δεδομένη. Και αν δεν καταφέρουμε γρήγορα να κλείσουμε τη συμφωνία, ας ψηφίσουμε, εν πάση περιπτώσει, να τελειώνουμε και έχει ενδιαφέρον να δει κανείς την γαλλική αντιπροσωπεία. Είναι δύσκολο να είναι κανείς στο Υπουργείο Εξωτερικού Εμπορίου όταν πρέπει να παρακολουθεί τον πρόεδρό σου που τρέχει δεξιά και αριστερά στον κόσμο. Δεν θα ήθελα να εργάζομαι στο εξωτερικό εμπόριο της Γαλλίας σε αυτή τη φάση. Λοιπόν, από τους κοιόδης εισηγητές Κέλλα. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω το αν το ότι πήγε στο Βερολίνο ανήκει στα ταξίδια αυτά ανά τον κόσμο. Δεν ήξερα ότι ήσασταν Γαλλίδα, λέει ο πρόεδρος. Δεν είμαι Γαλλίδα, είμαι Ευρωπαία, λέει η κυρία Κέλλα. Σαν κοινοβούλιο εμείς θα πρέπει να εμείνουμε στις απόψεις μας ανεξάρτητα από το ποια νου θα περάσει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να υπερασπιστούμε την άποψη του Κοινοβουλίου και να στηρίξουμε τον Ντέιβιντ όσο περισσότερο μπορούμε. Κάποιος άλλος και όδης εισηγητής από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πράγματι χτες ε, είχε πάει ο Γάλλος πρόεδρος στη Γερμανία για τα ευρωπαϊκά συμφέροντα συζήτησαν και όχι για την πρόθεση των γαλλικών συμφερόντων. Εν πάση περιπτώσει, επαναλαμβάνω και εγώ αυτό που είπε ο Κρίστοφερ, δεν χρειάζεται να ξαναγίνει συζήτηση από την αρχή. Η θέση του Κοινοβουλίου εξεφάστη σαφώς και υπήρξε ίσως μια μικρή πλειοψηφία στη λήψη της απόφασης, αλλά ε, αυτό που θα συμφωνήσω είναι με την πρόταση να κλείσουμε το θέμα γρήγορα χωρίς να υποχωρήσουμε ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γιατί τα επιχειρήματα είναι μαζί μας, εισαγωγικά, μας δικαιώνουν. Πρέπει να υπερασπιστούμε λοιπόν την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα πρέπει να συνενέσουμε με τη διαδικασία όμως. περιμένοντας να υπάρξει μια τελική λύση. Ευχαριστώ. Κάποιο άλλο σχόλιο. Όχι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο. Δεν υπάρχουν πολλά να προσθέσει κανείς ε, στην παρουσίαση του θέματος από τον εισηγητή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιμένει την ε, δεύτερη ανάγνωση και ένα πιθανό τριμερή διάλογο που θα εξαρτηθεί βέβαια από την απόφαση τη δική σας. Όταν γίνουν αυτά εμείς θα μπορέσουμε να διευκολύνουμε πλέον την διαδικασία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ανακοινωθεί επίσημα προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εμείς ε, νομίζω οδεύουμε παράλληλα με τις θέσεις του Συμβουλίου, αυτές που ανακοινώθηκαν το Δεκέμβριο και δεχόμαστε και τις τεχνικές τροπολογίες. Ε, αποδέχεστε επίσης και τις προσπάθειες που γίνονται για ε, επίλυση λύσης Καλά λέει ο Πρόεδρος. Σε περιπτώσει θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό στην ψηφοφορία το απόγευμα. Ο χρονισμός έχει σημασία. Αν θα είναι Ιανουάριος του 14 ή Ιανουάριος του 16. Περνάω τώρα στο σημείο 5 να καλωσορίσω τον κύριο Ρίτσαρντ Μπρότον. Υπουργό Καινοτομία τη Ιρλανδική Δημοκρατία, εκπροσωπεί τον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου και θα αναφερθεί στις προτεραιότητε της Ιρλανδική Προεδρίας. Να καλωσορίσω τον κύριο Μπρούτον. Είχα την δυνατότητα να συζητήσω μαζί του τον μήνα Δεκέμβριο στο Δουβλίνο. Ήταν μια ιδιαίτερα, θα έλεγα, χρήσιμη συζήτηση και νομίζω ότι οι συναντήσεις με το Συμβούλιο πριν από την έναρξη της Προεδρίας της κάθε χώρας είναι κάτι το ιδιαίτερα χρήσιμο. Και Μπράτον, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Είναι μεγάλη τιμή που βρίσκομαι εδώ μαζί σας και σας απευθύνω το λόγο. Είναι καθοριστικός δημοκρατικός θεσμός στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και νομίζω ότι ο καθηγητής κύριος Μορέιρα έχει βοηθήσει τα μάλα στη διαμόρφωση της ατζέντα για το διεθνές εμπόριο. Είναι η 7 Προεδρία της Ιρλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλες αυτές τις δεκαετίες που είμαστε μέλη έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο τα θεσμικά όργανα διαβουλεύονται με τους ε, ε, μπλεκόμενους φορείς αλλά και με τους πολίτες. Και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερος γι' αυτό. Η Επιτροπή σας εξετάζει τα διεθνή εμπορικά θέματα και εκπληρώνει πλήρως το ρόλο του συνομοθέτη. Οφείλουμε να διαμορφώσουμε την ατζέντα για την εμπορική πολιτική, ώστε και για τους πολίτες και για τις επιχειρήσεις και για όλους να είναι το αποτέλεσμα καλύτερο. Έχουμε εμπορικού εταίρους σε τρίτες χώρες και στις λιγότερο αναπτυσσόμενες και λιγότερο αναπτυγμένες χώρες κυρίως. Θέλω να συνεργαστώ μαζί σας και για νομοθετικά θέματα και για τις εμπορικές συμφωνίες. Θα κερδίσουμε όλοι αν καταλάβουμε καλύτερα την προοπτική του ενός και του άλλου. Ως Ιρλανδική Προεδρία αναλαμβάνουμε τις ευθύνε μας σε δύσκολους καιρούς για το διεθνές εμπόριο και την οικονομική δραστηριότητα και την ανεργία. Ζούμε μια οικονομική κρίση πολύ μεγάλη και είναι ε, το κάτω μέρος του οικονομικού κύκλου. Το έχουμε πέσει πολύ χαμηλά συγκριτικά με τις τελευταίες δεκαετίες. Σταθερότητα λοιπόν, δουλειές και απασχόληση είναι το σλόγγαν της Προεδρίας μας. Ε, έτσι ώστε να ανταποκριθούμε στην πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και οι πολίτες. Πρέπει να σημειώσουμε πρώτο, να δώσουμε νέα ανάκαμψη στους πολίτες και στις κοινότητες. Οι επενδύσει και το εμπόριο θα μπορέσουν να διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο. Πρέπει να αυξηθεί το εμπόριο για να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Αυτό θα είναι καταλήτης για να αποκτήσουν οι πολίτες ελπίδα και εμπιστοσύνη ότι θα υπάρξουν καλύτερες προοπτικές και θα βελτιωθεί το μέλλον το δικό τους και των παιδιών τους. Μήνυμά μας είναι ότι η Ευρώπη είναι ανοιχτή ε, στις επιχειρήσεις και για τις επιχειρήσεις. Το ανοιχτό μας πνεύμα σημαίνει ότι οι υπόλοιποι θα συνεχίσουν να ερμηνεύουν την Ευρωπαϊκή Ένωση ως εταίρο ειλικρινή, αξιόπιστο, με συνέπεια, με συνοχή, παραγωγή με ανάπτυξη ε, των σωστών πολιτικών, έναν εταίρο ο οποίος θα υπερασπιστεί τα δικαιώματα και τις προσδοκίες των πολιτών και των επιχειρήσεων και θα υποχρεώσει και τις τρίτες χώρες να τηρήσουν τις δικές τους ε, δεσμεύσεις σε επίπεδο διμερών συμφωνιών. Ως προς τον αντίκτυπο των εμπορικών συμφωνιών, σήμερα 26 εκατομμύρια άνθρωποι απασχολούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα θέματα αυτά και το όφελος λοιπόν από όλες τις συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου ε, μας οδηγεί σε 2 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης επιπρόσθετα. Και έτσι θα συμβάλλουμε σημαντικά για να αντιμετωπίσουμε μία από τις μεγαλύτερες κοινωνικές μάστιγες που που μας πλήττουν σήμερα, που είναι δηλαδή η ανεργία. Σε πολλές χώρες οι εξαγωγές είναι η μόνη πηγή ανάπτυξης στη σημερινή οικονομία. Οι επιχειρηματίες μας λοιπόν έχουν τη δημιουργικότητα, την τεχνολογία, τη φιλοδοξία να διαχύσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα σε όλες τις γωνιές ε, του πλανήτη μας. Θα πρέπει να έχουν νέες ευκαιρίες για πρόσβαση σε νέες αγορές μέσω νέων εμπορικών συμφωνιών. Και αυτά είναι στη πρώτη θέση του καταλόγου των προτεραιοτήτων μας. Μιλήσατε κύριε ε, πρόεδρε, για τα ωφέλη μιας ε, συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και η παρουσία σας εδώ υπογραμμίζει το πόσο σημαντικό είναι το θέμα αυτό. Μετά από τις συστάσεις της ε, Ομάδας Εργασίας Υψηλού Επιπέδου ΕΕ και ΕΕ, θέλουμε να ενισχύσουμε την διατλαντική αγορά. Είναι μια αγορά πολύ καλά ενωμένη. Έχουμε μεγάλες ροέ εμπορίου και επενδύσεων, ωστόσο πολλά περισσότερα θα μπορούσαν να γίνουν. Θα οργανώσουμε λοιπόν ένα άτυπο συμβούλιο στο Δουβλίνο, στο οποίο προφανώς θα σας προσκαλέψουμε κύριε Πρόεδρε και ελπίζουμε να παραστείτε για τα θέματα αυτά. Πρέπει λοιπόν να κεφαλαιοποιήσουμε πάνω σε αυτά που έχουμε ήδη επιτύχει και να αξιοποιήσουμε πλήρως το δυναμικό της διατλαντικής οικονομικής και επιχειρηματικής σχέσης. Οικονομικής και επιχειρηματικής σχέσης. Είναι πολύ σημαντικό το δυναμικό αυτό, άρα μόνο επιτυχία μπορεί να γίνει. Θα εκπέμψουμε ένα ισχυρό μήνυμα ότι δηλαδή ακόμα και σε, και, καιρούς ε, οικονομικών δυσχεριών και η ευρωπαϊκή και η αμερικανική οικονομία θέλουν να προχωρήσουν προς τα εμπρός, ανοίγοντας τις αγορές και όχι κλείνοντας και προστατεύοντάς τις. Και αυτό θα είναι σαφές μήνυμα στους εταίρους μας και ολοκληρώνουμε και μία άλλη ιστορική συμφωνία ελευθερού εμπορίου με τον Καναδά, ένας πολύ σημαντικός εταίρος διατλαντικός Βεβαίω οι δασμοί είναι χαμηλοί, ωστόσο με την Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου θα έχουμε σημαντικά ωφέλη και θα αρθούν διάφοροι περιορισμοί και εμπόδια, τα τελευταία εμπόδια. Ελπίζω να λυθούν γρήγορα τα εκκρεμή ζητήματα και να καταλήξουμε σε συμφωνία λίγα συντόμω. Βεβαίω και με, με άλλε οικονομίε θα θέλαμε να εμβαθύνουμε τι ε, εμπορικέ και οικονομικέ μα σχέσει, εκτό από τη ΣΥΠΑ και τον Καναδά. Ελπίζω να ξεκινήσουμε τι διαπραγματεύσει με την Ιαπωνία λίγαν συντόμω. Αυτό θα είναι πολύ σημαντικό γιατί σε αυτή τη συζήτηση θα συμμετάσχουν ε, δύο οικονομίες παγκόσμιας σημασίας. Καλό θα ήταν να γίνει και πρόοδος στις ε, διαπραγματεύσεις με την Ινδία, όπου μια συμφωνία ελευθέρου εμπορίου θα ήταν ευεργετική για αμφότερα τα μέλη. Και σε αυτό το πλαίσιο ε, θα μας βοηθήσει η συμφωνία αυτή στις σχέσεις μας με τις υπόλοιπες χώρες της περιφέρειας αυτής, της περιοχής αυτής μπορούμε να αξιοποιήσουμε και να εμβαθύνουμε ε, τις δυνατότητες ε, στις σχέσεις μας με την Κίνα. Να προετοιμάσουμε το έδαφος για να έχουμε μία, ε, τις σωστές προϋποθέσεις για να έχουμε μία καθοριστική συμφωνία για την πρόσβαση στην αγορά με την Κίνα. Και βέβαια θα πρέπει να καλλιεργήσουμε τις σχέσεις και με τους ε, πιο κοντινούς μας γείτονες. Μολδοβία, Γεωργία, Αρμενία. Οι εμπορικέ διαπραγματεύσει με αυτές τις χώρες σημειώνουν πρόοδο και θα φτάσουν σε πολύ ε, προχωρημένο σημείο κατά τη διάρκεια τη Προεδρίας μας. Σίγουρα έχουμε ε, δυσκολίες με τις ε, μεταρρυθμίσεις από την Αραβική Άνοιξη. Νομίζω ότι με τις εμπορικές συμφωνίες μπορούν οι χώρες αυτές της Βορείου να επιταχύνουν το ρυθμό των δημοκρατικών τους μεταρρυθμίσεων και να επιτύχουν ακόμα μεγαλύτερη πολιτική σταθερότητα. Όταν ξεκινήσουν οι, συνομιλίες για την απελευθέρωση των εμπορικών ροών, οι εταίροι μας θα πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένοι και μπορούμε εμείς να τους βοηθήσουμε σε αυτό. Οι εμπορικές συμφωνίες με το Μαρό, οι εμπορικές συνομιλίες με το Μαρόκο θα μας οδηγήσουν σε μια νέα δυναμική σχέση με αυτόν τον τόσο σημαντικό μας εταίρο, καθώς επίσης και με τους άλλους. Οι χώρες της ε, Νοτιοανατολικής Ασίας είναι πολύ σημαντικές για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια οικονομική ε, ζώνη μεγάλης σημασίας και ελπίζουμε ότι το δίκτυο συμφωνιών ελευθέρου εμπορίου έχει ήδη δρομολογηθεί και μπορεί να επικταθεί με την προσχώρηση σε αυτό το δίκτυο και άλλων χωρών, όπως για παράδειγμα της Ταϊλάνδης. Αυτό θα ήταν σημαντικό, γιατί η οικονομία αυτή είναι μεγάλος εταίρος στην παγκόσμια ε, οικονομική και εμπορική αλυσίδα. Αλλά και οι πολυμερείς συμφωνίες είναι σημαντικές για την Ιρλανδική Προεδρία. Ο ΠΟΕ είναι αυτός που καθορίζει τους κανόνες στο διεθνό, διεθνές εμπόριο και έτσι οι αλυσίδες αξιών επιμηκύνονται και όλοι μπορούν να επωφεληθούν με τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα και με την εξειδίκευση που θα έχει ο καθένας. Άλλωστε, οι λιγότερο ανεπτυγμένε χώρες μπορούν να επωφεληθούν από το εμπόριο και να αξιοποιήσουν τις ε, σχέσεις και τις διασυνδέσεις μεταξύ των διαφόρων αγορών. Η διευκόλυνση ε, στη συμμετοχή ε, στο εμπόριο, η διευκόλυνση του εμπορίου θα είναι και το βασικό θέμα της Υπουργικής Διάσκεψης του ΠΟΕ φέτος και προς όφελος των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών. Οι πιο φτωχές χώρες χρειάζονται ε, να δοθεί νέα πνοή στην ατζέντα της Ντόχας και να λυθούν διάφορα ζητήματα ώστε να επιταχυνθεί ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης σε αυτές πολύ σημαντικές είναι οι ευκαιρίες που υπάρχουν με τη δραστηριότητα του ΠΟΕ στη Γενέβη. Γνωρίζουμε πόσο μπορούν οι υπηρεσίες και η απελευθέρωσή τους να ενισχύσει το διεθνές εμπόριο. Θα μας ωφελήσει ως οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενθαρρύνουμε τις διαπραγματεύσεις για τις υπηρεσίες. Η Ιρλανδική Προεδρία θα λειτουργήσει επικοδομητικά ώστε να προχωρήσουν τα θέματα των υπηρεσιών στη Γενέβη. Θα καταλήξουμε σε συμφωνία για την εντολή διαπραγμάτευσης στις αρχές του 2013, εν ώψη της έναρξης των διαπραγματεύσεων στη Γενέβη. Στρέφουμε τώρα σε κάποιους από τους νομοθετικούς φακέλους που είναι εξίσου σημαντικοί. Προστασία των επενδύσεων απαραίτητο αναπόσπαστο τμήμα μιας εμπορική πολιτικής. Σημαντικό εργαλείο για να διευκολυνθεί η προστασία των επενδύσεων είναι κάτι που έχετε συμπεριλάβει στην ημερήσια σα διάταξη. Και ως Ιρλανδική Προεδρία θα συνεργαστούμε με εσά για την επίτευξη πολιτική συμφωνίας για ένα νομοθετικό πλαίσιο ώστε να έχουμε τη σωστή εξέλιξη στις, την επίλυση των διαφορών ως προς τις επενδύσεις και την προστασία αυτών και ούτω καθεξής. Μιλούμε και για τις άμεσες ε, ξένες επενδύσεις, οι οποίες έχουν μετά τις συνθήκες της Λαβώνας μπει ε, στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, πρέπει να καλύψουμε αυτό το κενό, να έχουμε νομική ασφάλεια, ώστε να έχουμε συμφωνίες που θα προστατεύσουν τους επενδυτές θα ολοκληρωθούν οι συμφωνίες με ισχυρή επενδυτική συνιστόσα, μεγάλο επενδυτικό σκέλος της συμφωνίας με, την Καναδά, τη Σιγκαπούρη, με τον Καναδά, τη Σιγκαπούρη, ενδεχομένως την Ιαπωνία, την Ινδία, άλλους σημαντικούς εταίρους και έτσι θα καλλιεργήσουμε ακόμα περισσότερο τη σχέση μας με την Κίνα όλο και πιο περίπλοκη είναι η ευρωπαϊκή νομοθεσία, αυτό είναι σαφές, ε, και τα πράγματα καθίστανται πιο περίπλοκα με τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δύο προτάσεις Omnibus υφίστανται και θέλουμε εμείς να τις προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο, να έχουμε ένα διάλογο με νόημα, επικοδομητικό ε, σε αυτούς τους φακέλους για να ε, καταλήξουμε σε συμφωνία κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας. Ως προς τις δημόσιες αγορές ή τις κρατικές προμήθειες, εμείς είμαστε ανοιχτοί σε νέες ιδέες. Πέρσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε μια πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για ένα νέο εργαλείο για τις ε, δημόσιες προμήθειες για να βελτιωθεί η πρόσβαση των ευρωπαϊκών εταιριών σε αυτή την αγορά των τρίτων χωρών. Ορισμένες αγορές για ε, δημόσιες συμβάσεις μπορεί να είναι πολύ ευρειέ και ένα εξαγωγέ να χάνει την ευκαιρία. Το Συμβούλιο εξετάζει αυτή τη στιγμή αυτή την πρόταση και θα έχετε μια δεύτερη ανταλλαγή απόψεων για αυτό το θέμα ε, σήμερα κάποια στιγμή αργότερα. Ως προς την νομοθεσία την εφαρμοστική, η σχετική ομάδα εργασίας του Συμβουλίου δουλεύει πάνω στην πρόταση της Επιτροπής για τη θέση σε ισχύ των διεθνών κανόνων για το διεθνές εμπόριο και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιλύσει γρήγορα, να καταρρύψει γρήγορα τα εμπορικά εμπόδια ε, στη σχέση της και με τις τρίτες χώρες που την ενδιαφέρουν. Ως προς τον κανονισμό για την πρόσβαση στις αγορές, το εμπόριο και η ανάπτυξη είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους, άρρηκτα συνδεδεμένα, προς όφελος και των ε, λιγότερων ανεπτυγμένων χωρών, αλλά και ημών. Για να έχουμε ευημερία στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες θα πρέπει να συντάξουμε συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης, τις οποίες ήδη διαπραγματευόμαστε. Θα πρέπει να τις ολοκληρώσουμε και να τις εφαρμόσουμε. Έτσι θα τις ωφελήσουμε. Θα σημειώσουμε πρόοδο και στον κανονισμό για την πρόσβαση στις αγορές. Είμαστε στο δεύτερο στάδιο. Έχει ήδη ξεκινήσει αυτό. Και θέλουμε να ε, συνεργαστούμε στενά μαζί σας για την ε, επίτευξη συμφωνίας σε δεύτερη ανάγνωση. Από τη στιγμή που μιλούμε για ανάπτυξη, θα ήθελα σε αυτό το στάδιο να αναφέρω τις σημαντικές αλλαγές ε, που έχουν γίνει στη Βερμανία Μιανμάρ. Η χώρα αυτή ήρθε, είχε σημαντικό μειονέκτημα και δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει το πολύ σημαντικό της δυναμικό λόγω των πολιτικών εξελίξεων όπως γνωρίζετε όλοι και ελπίζω γρήγορα να Εξετάσε την πρόταση να ξαναμπεί η Μιανμάρ Βιαρμία στο σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων για να αποκατασταθούν ε, τα προβλήματα και να ε, έχουμε τις γενικευμένες εμπορικές προτιμήσεις με την χώρα αυτή, ώστε να μπορέσει να ξαναμπεί στο δρόμο της ανάκαμψης και της, ανάκαμψης ανάπτυξης. Κύριε Πρόεδρε, οι ευθύνε μας είναι κοινέ, ημών και ημών. Ε, θέλουμε όλοι να στηρίξουμε την οικονομική ανάκαμψη, την ε, δημιουργία θέσεων επασχόληση. Θα είναι μεγάλη χαρά για μένα να συνεργαστώ στενά με όλου εσά του επόμενου έξι μήνες για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε όλες τις ευκαιρίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την εκτεταμένη επισκόπηση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι προτεραιότητες ε, της ε, Ιρλανδικής Προεδρίας παρουσιάστηκαν. Ευχαριστώ που μου ε, δώσατε μια δημόσια πρόσκληση για την συνάντηση στο Δουβλίνο. Θα ήταν μεγάλη μου χαρά να έρθω. Είναι πολύ σημαντικό να έχετε μια τέτοια πρόσκληση από το Συμβούλιο είναι άλλος ένας νέος τρόπος ε, να καταθέσει η Επιτροπή μας τις απόψεις της στο Συμβούλιο. Να καλωσορίσω και τους υπόλοιπους της Ιρλανδικής Αντιπροσωπείας, την κυρία Λόρεν Μπένσον και τον κύριο Τζέραλτ Μάμπς, μέλος ε, του Ιρλανδικού της GPC. Σας καλωσορίζω. Ο Ντανιέλ Κασπάρη από το ΕΠΠ. κύριε Υπουργέ, από το ΕΛΚΟ, Ντανιέλ Κασπάρη. Ε, καταλαβαίνετε γερμανικά, όχι. Ωραία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που είστε μαζί μας σήμερα για να μιλήσουμε για τα ε, σχέδιά σας. Ε, είναι τρία τα θέματα που με αφορούν. Το ένα είναι τα διατελαντικά ε, σχέδια που είναι κάτι που ενδιαφέρει πολύ την ομάδα μας όπως φάνηκε τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες, είμαστε έτοιμοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβουμε αποφάσεις ε, και να πάμε στον δρόμο των Αμερικανών ε, και χαίρομαι ιδιαίτερα που υπάρχει συνομιλία με τους Αμερικάνους έτσι ώστε όλοι στην Ευρώπη τελικά να δεσμευτούν για την επιτυχία αυτού του προγράμματος. Ε, θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί έχουμε τα δύο μεγάλα μπλοκ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ΣΥΠΑ που πραγματικά αν συνεργαστούν και αν είναι αυτό κομμάτι των προτεραιοτήτων σας θα αλλάξει ο κόσμος. Το δεύτερο θέμα είναι ε, το θέμα της ε, προστασίας των επενδύσεων. Δεν θέλω να μπω πολύ σε λεπτομέρειες, αλλά ανησυχώ ότι σε αυτό το θέμα θα ξαναζήσουμε αυτό που συνέβη σε κάποια κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η συζήτηση για το τι, ποιες είναι οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και ποιες όχι. Υπάρχει μια έρευνα για αυτό το θέμα και βλέπω ότι υπάρχουν και διάφορες τροπολογίες που κατατίθενται στο Κοινοβούλιο από διάφορα κράτη-μέλη και πραγματικά με ανησυχεί ειδικά το γεγονός ότι η κοινή εξωτερική πολιτική ε, μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας δεν θα είναι πραγματικά κοινή. Και πραγματικά στις ομάδες εργασία ε, του Συμβουλίου θα ήθελα να σας ζητήσω να υπάρχει ε, μια δράση ώστε να σταματήσει αυτή η αντιδραστική συμπεριφορά, γιατί πραγματικά θέλουμε από κοινού να έχουμε μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική εμπορίου. Πραγματική μάλλον πολιτική. Το τρίτο θέμα είναι οι κανόνες. Πραγματικά χαίρομαι που από κοινού σκεφτόμαστε για το πώς ε, θα καταφέρουμε μέσα από πρωτοβουλίες η Ευρωπαϊκή Ένωση να φροντίσει ώστε να τηρούνται οι κανόνες. Η Ρωσία ήδη από τον Αύγουστο έχει δείξει ότι δεν θέλει να τηρήσει πολλές ε, δεσμεύσεις. Ε, υπάρχει το dumping από την Κίνα. Αυτά είναι προβλήματα που πραγματικά πρέπει να σας θυμίσω. Και ξεκάθαρα θα ήθελα να μην πέσουμε σε προστατευτισμό. Θα ήταν λάθος αντίδραση. Θα πρέπει να σκεφτούμε έξυπνα ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ένα σωστό εταίρος, αλλά και όλοι να τηρούν τις, τους κανόνες. Πρέπει να είμαστε στεναρεί σε αυτή την ε, θέση, ε, γιατί η οικονομία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως παίζει και στη Ρωσία και στην Κίνα και σε άλλες τέτοιες ε, χώρες και θα είναι πολύ σημαντικό να εφαρμόσουμε εκεί τα συμφέροντά μας και θα είναι δύσκολο αν δεν τηρούνται οι κανόνες. Η εφαρμογή λοιπόν των κανόνων που από κοινού συμφωνήσαμε από τη στιγμή που είμαστε μέλη του ΠΟΕ, ε, πραγματικά θα πρέπει να τηρούμε τους κανόνες ε, και να μην κάνουμε ό,τι έκανε η Ρωσία τον Αύγουστο, γιατί τελείως θα πρέπει να πέσουμε σε προστατευτισμό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Πριν δώσω τον λόγο στον επόμενο μιλητή, να επαναλάβω αυτό που είπε ο Ντανιέλ Κασπάρη για τη νομική βάση των συμφωνήσεων. Αυτή είναι μια αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης μέσα από την κοινοτική μέθοδο. Δεν πρέπει τεχνικά να αλλάξει και να γίνει μεικτή συμφωνία όπως ε, κάποια κράτη-μέλη προσπαθούν να κάνουν. Οι συμφωνίες εμπορίου να γίνουν μεικτές εμπορίες. Αυτό θα είναι κάτι που πραγματικά θα προσπαθήσουμε να πατάξουμε και θα πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρη αντίδραση από την Ιρλανδική Προεδρία προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα από τους σοσιαλδημοκράτες, ο Ζόρς Κούτας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, να καλωσορίσω τον κύριο Μπάρτον στην Επιτροπή μας, εκ μέρους της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Να πω ότι με εντυπωσίασε το φιλόδοξο σχέδιό σας και να σας δώσω μια συμφουλή. Προσπαθήστε να επικεντρωθείτε όχι σε πάρα πολλούς ε, στόχους, γιατί είναι σημαντικό μετά από έξι μήνες τελικά να έχουμε αυτά αποτελέσματα. Και εγώ λίγο πολύ θεωρώ ότι η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών με την ΣΥΠΑ και τον Καναδά είναι το πιο σημαντικό, γιατί έχετε καλές ε, σχέσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Συμφωνώ πλήρως μαζί σας ότι πρέπει να έχουμε νέα πρόσβαση στην αγορά, νέες ε, αγορές, να βρούμε ε, νέες λύσεις ε, για τις ευρωπαϊκές επενδύσεις και να εφαρμόσουμε και τους κανόνες τους εμπορικούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης για τις χώρες της Ασίας ήταν πολύ σημαντικά τα όσα είπατε εξαιτίας των εξελίξεων σε επίπεδο ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια. Είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση σε αυτές τις χώρες και να σας το πω για ενημέρωση γιατί ήμουν πρόεδρος σε μια αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πέρυσι στο Λαός σε μια ε, συνάντηση ΑΚΕΠ που είναι η κοινοβουλευτική ε, διάσταση των ε, συνεδριάσεων ε, ΑΣΕΜ, ΑΣΕΑΝ. οι εταίροι από την ΑΣΕΑΝ ρωτούν πού θα είναι η επόμενη συνάντηση της ΑΚΕΠ το 2014. Η Ιταλία είχε πει ότι θα είναι αυτή που θα φιλοξενήσει, τελικά δεν θα το κάνει και η μόνη λύση ήταν να τους ενημερώσω τι θα γίνει στην Ευρώπη. Πού ακριβώς ε, δεν ξέρω. Ε, θα ενημερώσω τον Πρόεδρο, τον κύριο Σούλτς, ε, γιατί είναι μια καλή ευκαιρία για το Κοινοβούλιο. Και είναι μια καλή ευκαιρία και για σας να βρείτε μια λύση γιατί το 2014 είναι κοντά και θα μπορεί να βρεθεί λύση στο Συμβούλιο, γιατί θα έχετε... στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θα ήθελα λοιπόν να σας θέσω και ένα άλλο θέμα όσον αφορά στη συμφωνία με το Ουσμπεκιστάν. Ήμουν ο εισηγητής και γι' αυτό το θέμα. Το 2011 είχαμε αυτό το θέμα. Τότε δεν συνενέσαμε γιατί ήταν μια επέκταση στο κείμενο εξαιτία ε, ε, των ανησυχιών που είχαμε για την παιδική εργασία στη χώρα αυτή. Μετά το Κοινοβούλιο ψήφισε μια ενδιάμεση έκθεση και ζητήσαμε από το Ουσμπεκιστάν επισήμως να αποδεχτεί ε, κάποιες αποστολές του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας. Δεν το δέχτηκαν και αυτή τη στιγμή έχουμε κολλήσει. Δεν κινείται τίποτα. Ο πρόεδρος Μορέα, Μορέιρα έστειλε μια επιστολή στις αρχές, στο Συμβούλιο. Δεν κινείται τίποτα όμως. Νομίζω ότι δεν θα είναι καλό για μας ε, να έχουμε μια τελική ψηφοφορία που θα είναι αρνητική, γιατί έρχεται για το 2013 η επόμενη φάση και στην αρχή του χρόνου ήδη οι αποστολές του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας δεν θα ε, βρουν λύση σε αυτό το θέμα. Σας εύχομαι λοιπόν καλή τύχη τις προτεραιότητές σας ε, και είμαι αισιόδοξο για τις δυνατότητές σας, οπότε θεωρώ ότι θα έχετε καλά αποτελέσματα. Επόμενος, εκ μέρους των φιλελευθέρων, ο κύριος Καζάκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω από πλευρά τη δική μου πολιτική ομάδα των φιλελευθέρων δημοκρατών. Να σας συγχαρώ για την αποφασιστικότητα που επιδεικνύεται ελπίζω να εξελιχθεί σωστά η εξωτερική πολιτική στον τομέα τον εμπορικό και να προωθηθούν οι προτεραιότητες, στις οποίες έχουμε ήδη αναφερθεί. Δύο ερωτήσεις θέλω να σας θέσω. Η πρώτη. Κατάληξη των διαπραγματεύσεων με τη Σιγκαπούρη. Ξέρετε ότι το θέμα των κανόνων προέλευσης των προϊόντων ε, σαν μια μικρή οικονομία η Σιγκαπούρη έχει περιορισμένους πόρους και επεξεργάζεται πολλά προϊόντα τα οποία ίδια εξάγει σε γειτονικέ χώρες όπως η Ινδονησία, η Μαλαισία κτλ. Πώς μπορεί η Ιρλανδική Προεδρία ε, να μας διαβεβαιώσει ότι η παραγωγή σε άλλες χώρες του ΑΣΕΑΝ δεν θα εκμεταλλευτούν την ε, συμφωνία με τη Σιγκαπούρη. Γιατί στο παρελθόν ξέρουμε ότι τέτοιου είδους συμφωνίες έχουν χρησιμοποιηθεί παράνομα από άλλες χώρες της περιοχής που θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν τη συμφωνία αυτή. Είμαι επίσης συγητής για την ε, Ιαπωνία, τη συμφωνία με την Ιαπωνία. Μπορείτε να μας πείτε πού βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις με την Ιαπωνία. Ξέρω ότι τα NTB είναι ένα εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη αυτής της εταιρική συμφωνίας με την ε, Ιαπωνία. Υπάρχει τρόπος να πείσουμε τους Ιάπωνες να φανούν λιγότερο προστατευτικοί στις διαπραγματεύσεις αυτές. Και αν θα μπορέσουν με κάποιο τρόπο να απομακρύνουν αυτά τα εμπόδια, τα προστατευτικά, τα επόμενα χρόνια. Η τελευταία ερώτηση συνδέεται με τις προσπάθειες που κάνουμε από κοινού με το Συμβούλιο και την Επιτροπή να καταλήξουμε σε μία λύση για την μικροχρηματοδοτική βοήθεια. Ξέρουμε τη σημασία που έχει αυτή η βοήθεια για τις χώρες οι οποίες περιμένουν η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα. Υπάρχουν ε, διαφορετικές αντιλήψεις μερικές φορές και σε θέματα αρχής με το Συμβούλιο εδώ έχουμε διαφορές ε, και σε σχέση με τις εφαρμοστικές πράξεις και σε σχέση με τις κατεξουσιοδότηση πράξεις. Θα θέλαμε να υπολογίζουμε στην συνεργασία σας για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες αυτές που έχουμε με το Συμβούλιο. Ελπίζω λοιπόν κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας να σημειωθεί πρόοδος και σε αυτό το ντοσιέ. Ευχαριστώ. Κυρία Κέλλα από τους Πασίνους. Ευχαριστώ Υπουργέ που ήρθατε εδώ και μας εκθέσατε τις προτεραιότητες της Ιρλανδικής Προεδρίας. Κάποιες ερωτήσεις για σας. Σχέσεις με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Βλέπουμε ότι επιτέλους έχουμε ένα ενιαίο συμβούλιο και θέλει να ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία με τη ΣΥΠΑ. Η άποψή σας είναι ότι η ενότητα αυτή θα συνεχιστεί όταν περάσουμε στα συγκεκριμένα επιμέρους θέματα. Και εδώ τίθεται το θέμα της ε, συμπερίληψης της γεωργίας. Τι ενότητα μπορεί να έχει το Συμβούλιο γύρω από τα θέματα της Γεωργίας στα πλαίσια της συμφωνίας αυτής. Αναφέρθηκαν κάποιοι και στο γύρο της Ντόχα. Αυτό είναι χαρακτηριστικό της πολυμερούς αντίληψης, αλλά από την άλλη η συμφωνία με τη ΣΥΠΑ θα χρησιμοποιηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο και θα χρησιμοποιηθεί σαν υπόδειγμα και για άλλους μήπως είναι κάτι το οποίο απειλεί την πολυμερή αντιμετώπιση των προβλημάτων ε, των εμπορικών σε παγκόσμιο επίπεδο αυτού του είδους η δίμερης ανάμεσα σε δύο μεγάλα μπλοκ διαπραγματεύσεις. Τώρα για τον Καναδά. Ελπίζω τα εμπόδια να ε, ξεπεραστούν γρήγορα. τι γίνεται με το βόρειο κρέας και η Ιρλανδία είναι παραγωγός χώρα μεγάλη. Πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει μια πιθανή ε, σύγκρουση εδώ ανάμεσα στα Ιρλανδικά συμφέροντα και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα. Και ένα τελευταίο θέμα είναι η Ινδία. Είπατε ότι θα αναζητήσετε την πρόοδο ελπίζουμε να υπάρξει μια συμφωνία την Άνοιξη πριν από τις επερχόμενες εκλογές στην Ινδία. Αυτό το οποίο επιθυμεί η Ινδία, αν καταλαβαίνω καλά, είναι η δυνατότητα σχετική ελεύθερης διακίνησης των προσώπων. Ενώ ανάμεσα στα κράτη-μέλη υπάρχει μια, θα έλεγα, υπάρχουν διαφωνίες για το πόσο μπορούμε να δεχτούμε κάτι τέτοιο. Το Ηνωμένο Βασίλειο, σαν παράδειγμα, δέχεται ένα υψηλό ποσοστό ε, διακίνηση συνδών ε, πολιτών. Η Ινδία σκέφτεται επίσης και το θέμα της προστασίας των επενδύσεων. Αναφερθήκατε εσείς ότι το θέμα αυτό για σας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και η Αυστραλία ε, προσπαθεί να το εξαιρέσει από εμπορικές συμφωνίες και το ίδιο θέλει να κάνει και η Νότιος Αφρική και η κυβέρνηση της Ινδίας είπε ότι το θέμα αυτό δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται σε εμπορικές συμφωνίες. Πιστεύετε ότι αυτό καθιστά την εμπορική συμφωνία με την Ινδία ανέφικτη ή πιστεύει και το Συμβούλιο ότι το θέμα αυτό της προστασίας των επενδύσεων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και στις συμφωνίες με τον Καναδά και γενικότερα σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες γιατί όπως είπα είναι πάρα πολλές οι χώρες οι οποίες ανησυχούν ιδιαίτερα. Ευχαριστώ. Εκ μέρους τώρα της ΚΟΕ ο κύριος Πολ Μέρφη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την παρουσίασή σας. Σαφέστατα η Ιρλανδική κυβέρνηση και η Ιρλανδική Προεδρία έχουν ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο για το ελεύθερο εμπόριο Κάποιες ερωτήσεις θέλω να κάνω για αυτές τις συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου ως προς την απόφαση και την ε, ερώτηση της Σκάι Κέλλερ. Μία πρόσφατη υπόθεση ε, είχε αναλυφθεί από το Μηχανισμό Επίλυσης Διαφορών της ΝΑΦΤΑ ε, θέτης αμφισβητεί μία απαγόρευση του φράκιν ε, αυτό είναι ε, παράβαση των ελάχιστων προτύπων και είναι κατά παραβάση των ε, δικαιωμάτων απαλωτρίωσης. Ε, ως προς το φράκιν λοιπόν, είναι ένα πρόβλημα για τον δραυλικό κατακαιρματισμό στο σχιστολιθικό φυσικό αέριο, νομίζω ότι είναι αυτό. έχει σχέση και με τους επενδυτές στην Ιρλανδία θα πρέπει να υπάρχουν μέτρα μη διακρίσεων. Είναι πολύ μεγάλες ε, προκλήσεις αυτές και δεν μπορούμε να έχουμε τέτοιες προκλήσεις και από τις ε, καναδικές επιχειρήσεις. Δηλαδή να είναι ίση η όρη για όλους τους επενδυτές. Ε, δίδεται στη κυβέρνηση του Καναδά η δυνατότητα να ε, νομοθετήσει υπέρ του περιβάλλοντος, υπέρ του όποιου νομίζει, αρκεί να μην υπάρχει διάκριση αναλόγως με την προέλευση του εκάστοτε επενδυτή ή επιχείρησης. Θα πρέπει λοιπόν η Ιρλανδική η ιρλανδικη επιροεδρια να στηρίξει αυτή την ε, υπόθεση, να στηρίξει ε, την απόσυρση των επενδυτών από αυτό το μηχανισμό επίλυσης διαφορών της ΝΑΦΤΑ. Από εκεί και πέρα γνωρίζετε τις πολλές επικρίσεις από μη κυβερνητικέ οργανώσεις, ε, ε, συνδικάτα, μέλη Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται ούτως ή άλλως οι εμπορικέ διαπραγματεύσεις υπό πλήρη μυστικότητα με μεγάλη προτεραιότητα και πρόσβαση ε, για τους μέγαλο επιχειρηματίες αλλά καθόλου ε, για όσους εκπροσωπούν ε, τους εργαζόμενους και το καθεξής. Πώς τοποθετήσετε ως Προεδρία, πώς θα εμπλακεί στη διαδικασία αυτή η οργανωμένη κοινωνία των πολιτών σε σχέση με την συμφωνία με τη ΣΥΠΑ. Το Κοινοβούλιο θα δει την εντολή για τις διαπραγματεύσεις και πιο συγκεκριμένα για τη συμφωνία με τη ΣΥΠΑ. Σίγουρα υπάρχει απόκληση μεταξύ της θέσης Κοινοβουλίου και κυβέρνησης των ΗΠΑ ως προς την προστασία των δεδομένων και τα δικαιώματα ε, ιδιοκτησίας στα διεθνή ε, ε, με την ε, συμφωνία SWIFT, με την απόρριψη του ΆΚΤΑ που εμείς έχουμε ψηφίσει ως Κοινοβούλιο. Πολύ μεγάλες διαφορές λοιπόν μεταξύ Κοινοβουλίου και ήπα, Πώς θα, ε, πώς θα προστατευτεί η θέση του Κοινοβουλίου στις διαπραγματεύσεις με τη ΔΙΣΥΠΑ. Ε, και τρίτον, ως προς την Ινδία, έχετε σημειώσει πρόοδο σε σχέση με, το, με την αηφορία και τη βιωσιμότητα αυτό το σκέλος έγιναν ε, πολύ μεγάλες ε, ε, διαμαρτυρίες εναντίον των άμεσων ξένων επενδύσεων, διαδηλώσεις. αυτό δεν σας κάνει να αμφισβητείτε τι πολιτική θέλουμε να εφαρμόσουμε σε Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ινδία. Από εκεί και πέρα, στο Συμβούλιο έχουν συζητηθεί οι γραμμές γραμμέ για να υπάρχει σήμανση αγαθών που προέρχονται από του παράνομου απικισμούς των Ισραηλινών. Ε, πώς θα το προωθήσετε το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ολοκληρώνουμε αυτό τον πρώτο γύρο ερωτήσεων. Έχουν ζητήσει και άλλοι το λόγο. Πάρα πολλές ερωτήσεις, κύριε Υπουργέ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ για, τα, για το ενδιαφέρον σας και τις ερωτήσεις σας. για τον κύριο Κασπάρη. Αναγνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει προσπάθειες για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Περιμένουμε τώρα για την έκθεση της ομάδας υψηλού επίπεδου που θα λειτουργήσει έτσι ώστε να εκινήσουν οι διαδικασίες γρήγορα. Έχουμε κάποιες δυνατότητες προς όφελος και των δύο πλευρών. Ελπίζω όπως είπα να υπάρξει γρήγορη πρόοδος. Οργανώνουμε εμείς ε, μια ανεπίσημη συνάντηση με τον στόχο αυτό και σε καμία περίπτωση δεν διστάζουμε σαν Ιρλανδική Προεδρία εφόσον υπάρχει επιθυμία και από τις δύο πλευρές να προχωρήσουμε και ελπίζω ότι υπάρχει θα προχωρήσουμε. Αναγνωρίζω ότι για το θέμα της προστασίας των επενδύσεων ότι πρόκειται για έναν τομέα ο οποίος είναι τομέας αρμοδιότητας ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα προσπαθήσω να συνεργαστώ στενά λοιπόν με το Κοινοβούλιο, έτσι ώστε να αναγνωριστεί πλήρως η αρμοδιότητα αυτή και να τηρηθούν οι δεσμεύσεις. Το Συμβούλιο συνειδητοποιεί πλήρως της φάσης ε, ε, μη σεβασμού από πλευράς ορισμένων χωρών της αρχής αυτής και είναι, ε, είμαστε αποφασισμένοι να αντιμετωπίσουμε το θέμα γρήγορα. Για τον κύριο Κούτας, για τη συμβολή του να ασχοληθούμε με λίγα και σημαντικά και όχι με πάρα πολλούς στόχους ταυτόχρονα. Είναι πολύ σωστή η πρόταση, αυτή θα είναι η στάση που θα ακολουθήσουμε θα συγκεντρώσουμε την προσοχή μας σε τομείς τους οποίους μπορούμε να ε, σημειώσουμε πρόοδο και φυσικά η συμφωνία με τη ΣΥΠΑ είναι ο πρώτος και το στόχος μας. για το πότε θα γίνει το 14 η συνάντηση σε σχέση με το ΑΣΕΑΝ και αν μπορούμε να παίξουμε εμείς κάποιο ρόλο για να λύσουμε το πρακτικό αυτό θέμα θα προσπαθήσουμε. Αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες τις οποίες έχει θέσει το Κοινοβούλιο σε σχέση με το Ουσμπεκιστάν. Έχουμε πάρει κάποια μέτρα για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την αποτροπή της παιδικής εργασίας στη χώρα αυτή. Εμείς τα βήματα τα οποία κάνουμε λαμβάνουμε υπόψη τις αξίες της Ένωσης Προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε την παιδική απασχόληση. Σεβόμεθα τις κατευθυντήριες γραμμές και τις διεθνείς αρχές για την προστασία των παιδιών. Υιοθετήσαμε τις τελευταίες βασικές ρυθμίσεις για την, προστασία, την απαγόρευση της παιδικής απασχόλησης και ελπίζω ότι οι αρχές του Ουσμπεκιστάν θα συνεργαστούν με τους διεθνείς οργανισμούς και θα σεβαστούν τα δικαιώματα αυτά. θα ήταν ευκταίο, δεν θα ήταν ευκταίο το Κοινοβούλιο να σταματήσει τη διαδικασία αυτή. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ελέγχει απόλυτα έτσι κι αλλιώς η Προεδρία. Θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Τώρα για τα θέματα που έθεσαν οι φιλελεύθεροι. Σημείωσα αυτά τα οποία είπατε σε σχέση με τις ρήτρες στη συμφωνία με τη Σιγκαπούρη και τις ανησυχίες τις οποίες έχετε για το πόσο μπορεί να φανούμε εκτεθειμένοι με τις γειτονικές χώρες γύρω από αυτό. Για την Ιαπωνία υπάρχει ένας ξεκάθαρος οδικός χάρτης και υπάρχει εδώ ένα θέμα σε σχέση με, τις μύδα, με τα μη δασμολογικά τέλη. Ελπίζω να ξεπεράσουμε τη δυσκολία αυτή και θα θέσουμε ένα συγκεκριμένο χρόνο έτσι ώστε μέσα σε αυτό να προσπαθήσουμε να λύσουμε το θέμα για να απομακρυνθούν όλα αυτά τα εμπόδια τα οποία παρεμποδίζουν τις εμπορικές δυνατότητες που υπάρχουν για τη χρωματοδότηση. Συνειδητοποιώ τη σημασία που έχει το θέμα αυτό και σε σχέση με τις αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου και σε σχέση με τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου το θέμα έχει γίνει αντικείμενο συζήτηση επανειλημμένα. Ελπίζουμε οι δυσκολίες να ξεπεραστούν. Αν η Προεδρία μπορεί να βοηθήσει, φυσικά και θα το κάνει. Για την κυρία Κέλλα. Ξέρουμε ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές θα είναι έτσι και αλλιώς δύσκολες. Όπως και στην περίπτωση του Καναδά και των εμποδίων με τον Καναδά, όλα εξαρτώνται από την γενικότερη ισορροπία της συμφωνίας. Έτσι θα δούμε τα επιμέρους θέματα τα οποία μπορεί να τεθούν ειδικά για τη Γεωργία. Είναι αλήθεια ότι και το ξεκαθαρίσατε αυτό και προς τον Επίτροπο Δεγκούχτ ότι ο τομέας αυτός είναι ευαίσθητος για σας και οι ανησυχία σας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Και το τελικό αποτέλεσμα θα πρέπει σίγουρα να σέβεται και τις δικές σας ανησυχίες. Εγώ δεν νομίζω ότι η πιθανή υπογραφή και επιτυχία, εν πάση περιπτώσει, της πορείας για την υπογραφή της συμφωνίας με τη ΣΥΠΑ να είναι κάτι το οποίο θα υπονομεύσει την αντίληψη των πολυμερών εμπορικών σχέσεων. Όχι, θα είναι ένα κίνητρο θα τονίσει τη σημασία και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται. Δεν είναι αντιθετικές μεταξύ τους οι δύο αυτές ε, καταστάσεις. Σημείωσα και τις ανησυχίες σας για τις διαπραγματεύσεις με την Ινδία. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ ευαίσθητο και σε σχέση με τη διακίνηση των προσώπων και σε σχέση με το θέμα της προστασίας των επενδύσεων Ελπίζουμε, εν πάση περιπτώσει, το ταχύτερο δυνατό να καταλήξουμε σε μια ισορροπημένη λύση. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να ξεχωρίσουμε κάποια στοιχεία ήδη από τώρα τα οποία να αφαιρέσουμε από το σύνολο των διαπραγματεύσεων. Για τον κύριο Μέρφυ, Ιρλανδό συνάδελφο, τον ευχαριστώ για το ενδιαφέρον του και για τα καλά του λόγια. έθεσε αρκετά θέματα. Κάποια από αυτά με ξεπερνούν θα έλεγα σε επίπεδο ε, συνειδητοποίησης των λεπτομεριών τους. Συνειδητοποιώ την ανάγκη να προσπαθήσουμε να ισορροπήσουμε με τα θέματα προστασίας δημοσίου συμφέροντος το Κοινοβούλιο πράγματι θα πρέπει να πιστέψει ότι προσπαθούμε να ισορροπήσουμε τα συμφέροντα του κοινού από τη μία, των πολιτών δηλαδή και της βιομηχανίας και της οικονομίας από την άλλη. Η επιθυμία μας ακριβώς είναι να εξισορροπήσουμε ε, τα πράγματα αυτά. Έτσι μόνο θα μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντα αυτά με το σωστό τρόπο και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να κάνουμε στις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών στις σχέσεις με τις Ηνωμένε Πολιτείες έχουμε πράγματι πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά, έχουμε σημαντικές διαφορές μεταξύ μας, αλλά η δυσκολία ακριβώς των διαπραγματεύσεων είναι η προσπάθεια εξισορρόπησης των διαφορών χωρίς να αποκρύβουμε και να ε, αγνοούμε τις βασικές μας αρχές. Πρέπει να τις συζητάμε με ξεκάθαρο τρόπο, να αναζητούμε την πρόοδο, Και το βασικό είναι ότι από τις εμπορικές συμφωνίες και από τις εμπορικές δραστηριότητες γενικότερα ανάμεσα σε διάφορες χώρες και ομάδες χωρών ε, υπάρχουν ωφέλη και για τους δύο. Τώρα για την Ιαπωνία. Ξέρετε ότι υπάρχουν ορισμένα πολύ σημαντικά θέματα Και εσείς όπως είπατε πρέπει να υπάρξει μια κάποια ισορροπία σε σχέση με αυτό. Και για τα θέματα της, ε, της επισήμανσης των προϊόντων ή της ετικετοθεσίας στα προϊόντα είναι θέματα στα οποία δεν μπορώ να σας δώσω σε αυτή τη φάση απαντήσεις. Δεν είμαι αρκετά ενημέρος. Να δώσω το λόγο τώρα στους άλλους ομιλητές. Πριν το κάνω, ε, κάποιες ε, σκέψεις. Δεν διαπραγματεύεται το Συμβούλιο εξ ονόματος της Ένωσης. Ε, η Επιτροπή είναι αυτή που είναι υπόλογη για την Ένωση και στις, μπροστά μας και για τις διαπραγματεύσεις αυτές. Αλλά για να το κάνει αυτό θα πρέπει να γνωρίζει τις απόψεις του Συμβουλίου. Έχει σημασία λοιπόν η θέση του Συμβουλίου να αντικατοπτρίζουν τις κοινέ μας θέσεις και πώς το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα τροφοδοτήσουν την Επιτροπή έτσι ώστε να επηρεάσουν τις διαπραγματεύσεις. Η σχέση μας με το Συμβούλιο είναι διαφορετική λοιπόν από αυτήν με το Συμβούλιο. Η Επιτροπή είναι υπόλογος απέναντί μας, ενώ το Συμβούλιο λέει ο Πρόεδρος δεν είναι. Ο κ. Στάζνη για το ΕΛΚ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την αναρκτήρια ομιλία σας, με την οποία συμφωνώ και την υποστηρίζω. Συμφωνώ με τα σημεία στα οποία επικεντρωθήκατε κυρίως για την Αμερική, όχι μόνο γιατί είμαι ο εισηγητής για τον Καναδά Ελπίζω ότι θα χρησιμοποιήσετε την Ιρλανδική σας ιδιότητα και θα, φτάσετε, θα φέρετε σε πέρας ε, τις διαπραγματεύσεις, αλλά και επισήμως θα ανοίξετε τις ε, διαπραγματεύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης είπα. Γιατί αν όχι οι Ιρλανδοί, ποιος άλλος ε, μπορεί να το κάνει. πιο πολλοί Ιρλανδοί υπάρχουν εκεί παρά στην Ιρλανδία. Και πρέπει να υποφεληθούμε από αυτό. Γιατί το εμπόριο, όπως είπατε, Οφελεί και τις δύο πλευρές. Και αν έρθουμε πιο κοντά, όπως είπε και ο συνάδελφος Κασπάρη, υπάρχουν πολλές προ... προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Γιατί όσο πιο στενά συνεργαζόμαστε στον τομέα του εμπορίου, θα ε, υποφεληθούμε και εμείς και οι υπόλοιποι με την παγκόσμια σταθερότητα που θα επιφέρει η συμφωνία. Υπάρχουν πολλές ερωτήσεις για τον Καναδά και τη ΣΥΠΑ που θα αφήσω Μιλήσατε για την Σιγκαπούρη, την Ιαπωνία. Ήδη έχουμε μια συμφωνία με την Νότια Κορέα. Σε αυτή την περιοχή θέλω να σας ρωτήσω αν σχεδιάζετε ή αν πρόκειται να δώσετε έμφαση στην Ταϊβάν. Σε αυτό το κοινοβούλιο έχουν ήδη γίνει κάποιες δραστηριότητες ε, και ενδιαφέρεται ιδιαίτερα η Ταϊβάν και πραγματικά ε, για το μέγεθός της η χώρα είναι πολύ μεγάλη κινητήριος δύναμη στην περιοχή και θέλουν να απορροφήσουν ε, αγαθά και υπηρεσίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιμονούν. Και η ε, Ιρλανδία δίπλα από την μεγάλη αυτή αρκούδα, την Κίνα, όχι τη Ρωσία, την, το κινέζικο πάντα, θα μπορέσει να βοηθήσει. Ελπίζω λοιπόν να σκεφτείτε λίγο αυτά τα θέματα. Ο Χέλμουτ Σούλτς από την ΚΟΕ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον Υπουργό για, τις... για τα όσα μας παρουσίασε ε, σχετικά με τους στόχους της Ιρλανδικής ε, Προεδρίας. Ε, να πω κάτι ακόμα για την Τόχα και τον ΠΟΕ και για το σύστημα εμπορίας. Άκουσα ότι θέλετε να πάτε παραπέρα ε, στο θέμα του συστήματος ε, του πολυμερούς εμπορίου. Το θέμα είναι αν μπορεί το Συμβούλιο να πάει προς αυτή την κατεύθυνση, γνωρίζοντας τις δυσκολίες που έχουμε σε αυτόν τον τομέα, ειδικότερα στον τομέα της γεωργίας. Αν δείτε τα κεφάλαια για τη γεωργία και τα, τους διάφορους ε, φραγμούς που υπάρχουν στις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, πραγματικά αμφιβάλλω κατά πόσο θα είναι αυτό εύκολο. Αυτό που μπορεί να παρουσιάσει η Προεδρία στην Κομισιόν, θυμίζω τα λόγια του Προεδρού ότι η Κομισιόν είναι αυτή που διαπραγματεύεται, ε, θα μπορέσει να βοηθήσει ώστε να υπάρχει μια ριζοσπαστική αλλαγή σε αυτό τον τομέα. Η Αμερικανική Ήπειρος επίσης είναι ένας σημαντικός πυλώνας για τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών. Όταν μιλάμε για προτεραιότητες, λοιπόν, να πούμε ότι δεν είναι μόνο της Ιρλανδικής Προεδρίας ε, προτεραιότητα να προχωρήσει σε αυτό τον τομέα. Υπάρχουν ε, προσδοκίες ε, και από την Λατινική Αμερική για μια εμπορική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία οδήγησε σε κατάληξη των διαπραγματεύσεων με το Περού και την Κολομβία. Αυτό σημαίνει ότι αυτή την εποχή όπου ο πρόεδρος Μπαρόζο θα συμμετάσχει στη Χιλή, στην Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Λατινικής Αμερικής, θα υπάρχει ένα θέμα για την εμπορική πολιτική. Πώς θέλετε λοιπόν να αντιμετωπίσετε αυτές τις προσδοκίες σε πρώτη φάση της ε, ε, τριμερούς προεδρίας που ανήκει με τη δική σας προεδρία. Ήδη αναφέρθηκε η ΣΕΤΑ, η Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία, νομίζω ότι σχετίζεται με τα ε, κεφάλαια για την ε, προστασία των ε, επενδύσεων. Υπάρχουν πολλές αμφιβολίες σχετικά με τις ε, τους διακανονισμούς μεταξύ κρατών και επενδύσεων κρατών. Ε, θα έχετε μία θέση τέτοια ώστε με ειλικρινή τρόπο ε, να υπογραμμίσετε τη θέση του Κοινοβουλίου που είναι υπέρ της, του διακανονισμού μεταξύ κρατών. Δεν θέλουμε αυτό το κεφάλαιο να συνεχίσει προς την κατεύθυνση που το κοινό αυτή τη στιγμή αντιλαμβάνεται. Δηλαδή προς τον διακανονισμό ε, κράτους, ε, μεταξύ κράτους και επενδυτών. Αναφέρθηκε επίσης το θέμα της ε, πνευματικής ιδιοκτησίας. Η άκτα είναι ε, ένα θέμα που εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο. Τι θέλετε να κάνετε με την ολοένα ε, και αυξανόμενη ευαισθητοποίηση των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διανοητική διοκτησία είναι ένα από τα υπέρ της οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως χρειαζόμαστε κοινού κανόνες για να έχουμε μια συνεργασία που θα είναι αμοιβαίως υποφελής και θα επιλύει ζητήματα που αφορούν στην ανάπτυξη των οικονομιών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υπολείπων χωρών. Τι μπορεί να φέρει στο τραπέζι της Κομισιόν του Συμβούλιο ως προς αυτό το θέμα των ε, διαφωνιών και σχετικά με την άκτα. Ευχαριστώ. Και μια τελευταία ε, παρέμβαση από τον Ρόμπερτ ε, Στέρντι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μόλις ήρθα από την Επιτροπή Γεωργίας και υπάρχουν κάποιες τροπολογίες ε, στην πρόταση ε, ΑΣΑΠ. Και μιλάω ως ε, ένας ε, γεωργός που έχω έρθει πολλές φορές στην Ιρλανδία και θα ήθελα να ξεφορτωθούμε την κοινή αγροτική πολιτική, αλλά δεν με αγαπούν στην Επιτροπή μου για αυτά που λέω. Πίτερ, εξαίρετα τα σχόλιά σου Απλώς μπορείς να μας εξηγήσεις. Υπάρχει αυτή τη στιγμή διαπραγμάτευση μιας ε, συμφωνίας ε, συναλλαγών. Μόλις ε, τελειώσουν μπορούμε να πάμε σε μια συμφωνία με τη ΣΥΠΑ και τα περισσότερα θέματα έχουν να κάνουν με τη γεωργία, με το γαλακτικό οξύ στο κρέας, με τα γενετικά τροποποιημένα. Ε, ε, έχουμε κατά κάποιο τρόπο ε, δεχτεί ότι θα πρέπει να έχουμε γενετικά τροποποιημένα, τι θα είναι αυτό σόγια, δεν ξέρω. Αλλά αν λαμβάνουμε υπόψη μας πόσο σημαντική είναι η γεωργία για τους Ιρλανδούς, 108 δολάρια έξτρα πληρώνουν για τις γενετικές τροποποιημένες σόγες και εισάγουν και κρέας. Ελπίζω λοιπόν να τα δούμε λίγο πιο ευρέως τα θέματα αυτά. Γιατί ε, πρέπει να δούμε τι κερδίζουν οι οικονομίες αυτών των χωρών από τη Γεωργία. Είναι λίγο πιο ευρύ το θέμα και όλα αυτά πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε πριν γίνει η συμφωνία με τη ΣΥΠΑ. Συνήθως οι μικρές χώρες όπως η Ιρλανδία τα πάνε πολύ καλύτερα στις διαπραγματεύσεις από ότι οι μεγάλες. Οπότε αδειμονούμε να έχουμε καλά αποτελέσματα από τι διαπραγματεύσει σα. Αλλά θα ήθελα και τη δική σα γνώμη σχετικά με το τι θεωρείτε για τη γεωργία και αν θα έπρεπε, να δοθεί πολύ, αν θα έπρεπε ή όχι να δοθεί πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτό. Πόσες προπολογίες ακριβώς είπατε ότι έχουν υποβληθεί. 8.000. Ψηφίζουν για 9 ώρες. 9 ώρες θα κρατήσει η ψηφοφορία, λέει, εκτός μικροφώνου βέβαια. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι θα τελειώσουν αυτό το μήνα. Να δώσω το λόγο στον κύριο Υπουργό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ένα πολύ, μια πολύ απλή ερώτηση στον Υπουργό. Ποια είναι η άποψή σας για αυτό το οποίο εγώ ονομάζω ε, ή πολιτικοποίηση των εμπορικών συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πράγματι, πράγματα που έχουν γίνει πολύ χειρότερα από τότε που η συνθήκη της Λισαβόνας έδωσε στο Κοινοβούλιο το δικαίωμα της συναπόφασης. Λοιπόν, ο Πρόεδρος, η απουσία των θεμάτων το, για τη Μερκοσούρ στην ομιλία σας σημαίνει ότι το Συμβούλιο πλέον δεν δίνει προτεραιότητα στα θέματα αυτά. Αυτή είναι η δική μου ερώτηση ως πρόεδρος. Και τι περιμένετε να ε, προκύψει από τη συνάντηση στο Σαντιάκο της Χιλής μεταξύ των εκπροσώπων της Επιτροπής και των Υπουργών της Ζώνης του Μερκοσούρ. Δεν θα πρέπει να γίνει προσπάθεια να δοθεί νέα πνοή στις διαπραγματεύσεις. Ή μήπω πιστεύετε ότι είναι αυτές καταδικασμένες, δεν έχει νόημα να Από εκεί και πέρα, ε, πώς θα το, ή πώς περιμένετε ότι οι εταίροι μας της Μερκοσούρ έχουν την ευθύνη να δώσουν πνοή στις ε, διαπραγματεύσεις με τη Μερκοσούρ. Αυτά για τη Μερκοσούρ. Να σας ρωτήσω τώρα για την Ινδία. Πολλοί συνάδελφοι έθεσαν το θέμα της Ινδίας. Εγώ θα ήθελα να το θέσω κάπως διαφορετικά. Δηλαδή, είναι σαφ σαφής πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης η εξής. Οι εμπορικές συμφωνίες πρέπει να είναι φιλόδοξες, ευραίως πεδίου και σε μεγάλο βάθος. Δηλαδή, να όσο ε, τον περισσότερα θέματα εμπορικά, αγαθά, υπηρεσίες, δημόσιες αγορές, κρατικές προμήθειες, ε, επενδύσεις ε, κτλ. Και σε, όσο δεν το μεγαλύτερο βάθος, δηλαδή όσο δεν λιγότερα εμπόδια δασμολογικά και ούτω από ό,τι καταλαβαίνω, οι στόχοι μας αυτοί τίθενται εν κινδύνο στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Ινδία. Ε, ίσως γιατί δεν υπάρχει λύση στο, στο κεφάλαιο για την αηφόρο ανάπτυξη οι διαπραγματεύσεις με την Ινδία ενδεχομένω δεν θα πετύχουν αυτούς τους τρεις στόχους που έχουμε πάντοτε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. ώστε να τον πιο ευρύ πεδίο εφαρμογή και ώστε να το μεγαλύτερο βάθος ε, για την κατάρριψη των ε, εμπορικών και δασμολογικών ε, εμποδίων και ώστε να το μεγαλύτερη επίτευξη των στόχων της αηφόρου ανάπτυξης. Αυτά είναι τα τρία σκέλη που πάντοτε μας ενδιαφέρουν. Πιστεύετε ότι ως Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνουμε εξαίρεση για την Ινδία τα έχουμε στενότερο πεδίο εφαρμογή, ε, να μην έχουμε του στόχου αηφόρου ανάπτυξη, επειδή πρόκειται για την Ινδία. Ε, είναι ανησυχία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αυτή και χρειαζόμαστε τη γνώμη του Συμβουλίου, να ξέρουμε πώ τοποθετείται. Σε ποιο βαθμό μπορούμε να ασκήσουμε πίεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να το πετύχουμε αυτό που θέλουμε, δηλαδή οι εμπορικές μας σχέσεις στο μέλλον με την Ενδία να ευθυγραμμίζονται με το πρότυπο, με την οτροπία που έχουμε εν γέννη για τις εμπορικές μας συμφωνίες με τους υπολείπους μας εταίρους. Σας δίνω το λόγο κύριε Ποριέ. ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής σας για όλες αυτές τις ερωτήσεις που μου έθεσαν. Ο Πίτερ με ρώτησε εάν η Ιρλανδία είναι η καλύτερα τοποθετημένη χώρα, αν θέλετε, βρίσκεται στην πιο καλή θέση για τη συμφωνία με τη ΣΥΠΑ. Ξέρετε, ε, σε μη... ο Ιρλανδός ε, ήταν ο εκπρόσωπος του Αμερικανικού Πανεπιστημίου, ο οποίος ε, υπέγραφε μια συμφωνία για την έρευνα και ανάπτυξη μαζί με ένα Ιρλανδικό Πανεπιστήμιο στη ΣΥΠΑ προσφάτως, ενώ ο αντίστοιχος εκπρόσωπος του Ιρλανδικού ε, πανεπιστημίου ήταν Αμερικανός. Με αυτό απαντώ στο πόσο στενές είναι οι σχέσεις μας και πράγματι ε, μπορούμε να προχωρήσουμε τα θέματα με τη ΣΥΠΑ. Τώρα, ως προς την Ταϊβάν, ε, σίγουρα η ατζέντα είναι πολύ βεβαρημένη. Αλλά είναι πολλές οι δυνατότητες σε βάθος χρόνου. Πρέπει να τις αξιοποιήσουμε. Ο κύριος Σούλτς μίλησε για τη Λατινική Αμερική, το S&D. Σίγουρα είχαμε συμφωνίες με την Κολομβία, το Περού μεταξύ άλλων. Ε, πολλές συζητήσεις διεξάγονται αυτή τη στιγμή με τους εταίρους της Μερκοσούρ. Ο Επίτροπος Ντεκούχτ συμμετέχει ενεργά σε όλες αυτές τις διαπραγματεύσεις. Πράγματι ο ρυθμός είναι πιο επιβραδυμένος, πιο βραδύς από ό,τι περιμέναμε. Ε, διάφορες δυσκολίες υπάρχουν εκεί όμως ε, σίγουρα πάρα πολλές ευκαιρίες ε, προκύπτουν σε αυτή την ε, ταχαίως αναπτυσσόμενη περιοχή του πλανήτη μας. Το Συμβούλιο δεν έχει αποκλείσει τη δυνατότητα ύπαρξη πολλών ευκαιριών σε αυτή την Ήπειρο. Βραχυπρόθεσμα όμως τα ωφέλη δεν θα είναι τόσο ορατά, πιο, πιο μακροπρόθεσμα θα είναι ορατά και προχωρούν αυτά τα πράγματα αν όχι και με τόσο γρήγορο ρυθμό. Τώρα, ως προς την άκτα, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ε, ε αντιγραφής και το καθεξής, copyright, θα ήθελα να πω ότι όπου έχουμε πολιτική, πολιτική π.χ. για τη γεωργία, για το copyright, όλα αυτά ε, είναι, όταν έχουν ψηφιστεί και εγκριθεί και δεν αλλάζουν, ε, τα λαμβάνουμε υπόψη στις διαπραγματεύσεις με τους άλλους εταίρους μας. Ως προς το copyright όμως, σίγουρα πρέπει να καταλήξουμε και σε καλύτερη ισορροπία εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να μπορέσουμε να συμμετάσχουμε και καλύτερα να αξιοποιήσουμε καλύτερα τις ευκαιρίες της ψηφιακής οικονομίας. Εγώ λοιπόν θα απαντούσα ε, ναι, καταφατικά. Ε, είμαι και στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και νομίζω ότι ξεκινά πλέον η συζήτηση στην Ευρώπη για το ε, πώς θα πρέπει να μεταρρυθμίσουμε την νομοθεσία για το copyright και κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας τουλάχιστον ε, ελπίζουμε να ξεκινήσει η συζήτηση και να μπουν κάποιες βάσεις για τη συζήτηση. Πάρα πολλές είναι των ΜΕΝ και των ΔΕ. Πολύ δύσκολο το αντικείμενο αυτό, πολύ δύσκολο να εξορροπήσουμε τα συμφέροντα και οι χρήστες όμως και οι δημιουργοί διαδικτυακού περιεχομένου ε, ενδιαφέρονται και είναι προς το συμφέρον αμφωτέρων να επιτευχθεί συμφωνία για να έχουν όλοι όσο το περισσότερες ευκαιρίες. Είναι σημαντικό αυτό το πεδίο σίγουρα, όμως όταν μιλούμε για εμπορικές συμφωνίες δεν θέλουμε να είμαστε καινοτόμοι σε αυτό ακριβώς το σκέλος τους, π.χ. τη γεωργία ή το copyright. Εκεί διαπραγματευόμαστε βάσει της εντολής που μας έχει δοθεί. Επομένως, ε, θα σεβαστούμε την υφιστάμενη θέση ε, που έχει θετηθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια αυτών των διαπραγματεύσεων. Ο Πρόεδρος έθεσε το εξής θέμα. Μήπως οι, οι φιλοδοξίες μας έχουν ε, τεθεί στο περιθώριο ή έχει κατέβει αν θέλετε ο πύχης των ε, φιλοδοξιών μας ε, προκειμένου να πετύχουμε συμφωνία με την Ινδία. Θα έλεγα ότι πρόοδο σε διαπραγμάτευση σημειώνεται μόνο όταν υπάρχουν ευκαιρίες να βρεθεί μια κάποια συμφωνία. Και στην τελική η συμφωνία που προκύπτει εντάσσεται ε, στη δικαιοδοσία της συναπόφασης. Άρα, όταν επιτύχουμε μια συμφωνία, σε όποια σημεία και αν επιτύχουμε συμφωνία, θα μπορέσετε το Κοινοβούλιο να τοποθετηθείτε και να πείτε αν σας αρέσει και αν είναι αρκετά φιλόδοξη. Εμείς προσπαθούμε να αυξήσουμε τις πιθανότητες, να έχουμε όσο το περισσότερες ευκαιρίες για να πετύχουμε συμφωνία και ελπίζουμε ότι στο τέλος δεν θα είναι υπερβολικά ρηχή η συμφωνία αυτή αλλά πρέπει να δούμε πρώτα ποια μορφή θα πάρει, πώς ακριβώς θα διαμορφωθεί το κείμενο. Ο κύριος Ντάρτμουτ έθεσε κάποια θέματα που ε, είναι εκτός της αρμοδιότητάς μου, δεν είναι πολύ ε, καλά, ε, δεν, έχω εγώ τη δυνατότητα, την εξουσία να αναδιατυπώσω τη, συμφω... τη συνθήκη της Λισαβόνας. Σίγουρα οι εμπορικές μας συμφωνίες και συναλλαγές έχουν πολιτική χρειά, πάντοτε την είχαν, αυτό είναι λογικό. Ε, όταν ε, ε, κάθε έθνος επιθυμεί και παίρνει την απόφαση να ανοίξει την αγορά του, σίγουρα πρέπει να μεριμνήσει ώστε οι ευαισθησίες του λαού του να ληφθούν υπόψη. Νομίζω λοιπόν ότι αναθεωρούνται πάντοτε οι οικονομικές και εμπορικές μας πολιτικές αναλόγως με τις συμφωνίες μας και νομίζω ότι αυτό που καταφέραμε, δηλαδή ε, και το Συμβούλιο αλλά και το Κοινοβούλιο να μπορούν να διαμορφώνουν αυτές τις διαπραγματεύσεις και να δίνουν τις κατευθυντήριες γραμμές ή να τις επικυρώνουν είναι ε, ο σωστός τρόπος γιατί έτσι επιτυχάνουμε ισορροπία ε, καλύπτοντας ε, τις ανάγκες των πολιτών μας και πετυχαίνουμε να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη εμβάνθηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, με την πάροδο του χρόνου. Θα θυμάστε ότι ξεκινήσαμε με ένα-δύο βασικά προϊόντα, ενώ τώρα είμαστε πολύ πιο συνολικοί στις συμφωνίες μας αυτές. Σίγουρα υπάρχουν ωφέλη με το μοίρασμα της, με την εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας γιατί μια χώρα ατομικά δεν μπορεί να έχει την ίδια επιρροή στο παγκόσμιο στερέαμα, στο διεθνές στερέωμα. Ο κόσμος αλλάζει και πρέπει να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις με διαφορετικούς τρόπους πλέον, ε, με την έλευση και την εδραίωση της παγκοσμιοποίησης. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Να υπενθυμίσω ότι η βάση της συνθήκης Λισαβόνας είναι υποχρεωτικό η εξωτερική εσωτερικές, η πολιτική ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική της δράση πρέπει να παρουσιάζει συνέπεια και συνοχή. Δηλαδή, η εξωτερική πολιτική, η αναπτυξιακή πολιτική, η πολιτική για τις εξωτερικές εμπορικές σχέσεις είναι τρεις πολιτικές που πρέπει να παρουσιάζουν συνέπεια και συνοχή μεταξύ τους, αλλά και συνέπεια και συνοχή με τις εσωτερικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε σχέση με την εσωτερική της επικράτεια. Να σας ευχαριστήσω θερμά κύριε Υπουργέ. Είστε ευπρόσδεκτος ανα πάσα στιγμή στη δική μας Επιτροπή. Κάθε μέρα θα είστε ο εταίρος μας, ο συνεργάτης μας για τους επόμενους έξι μήνες. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Uh, λοιπόν, το επόμενο... Συνεργασία, λοιπόν, για τις πρόδρομες ουσίες στα ναρκωτικά με τρίτες χώρες. Τι, είναι τούτο, λέει ο πρόεδρος. Χημικές ουσίες, οι οποίες χρησιμοποιούνται συχνά για παράνομη ε, παρασκευή ναρκωτικών ουσιών Υπάρχουν ε, πολύ συγκεκριμένοι τρόποι εμπορία των ουσιών αυτών και υπάρχει μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διεύρυνση της εμβέλειας αυτών του κανονισμού για να συμπεριληφθεί η εφεδρίνη και η ψεύδο εφεδρίνη. Ε, medicines from which they can be rather easily extracted and used μπορούν να ε, πάρουν τις ουσίες αυτές ε, από τα φάρμακα που κυκλοφορούν με άδεια έτσι ώστε να παρασκευάσουν το ναρκωτικό ανάμεσα σε άλλα ε, την ναρκωτική ουσία αμφεταμίνη. Ο κύριος Προύστ είναι από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα εισηγητής. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αγαπητέ συνάδελφοι, η πρόταση κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως είπατε, τίνει στην αναθεώρηση της ε, εποπτείας της εμπορίας πρόδρομων ναρκωτικών ουσιών ανάμεσα στην κοινότητα και τις τρίτες χώρες. Θέλουμε να τροποποιήσουμε το πεδίο εφαρμογής του ισχύοντος κανονισμού, προσθέτοντας την εφεδρίνη και την εφεδρίνη. Η Επιτροπή θέλει να επωφεληθεί από την αλλαγή αυτή και για την προσαρμογή της επιτροπολογίας στη συνθήκη της Λισαβόνας. Οι πρόδρομες ουσίες είναι νόμιμες ουσίες που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή ζωή και που μπορεί να χρησιμοποιηθούν καταχρηστικά για συνθετικά ναρκωτικά. Είναι οι λεγόμενες πρόδρομες ουσίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα του κανονισμού. Τριών ειδών είναι οι κατηγορίες αυτές των προϊόντων. Η πρώτη κατηγορία ανήκει σε μια πολύ δεσμευτική, θα έλεγα, μορφή ελέγχου σε σχέση με τη 2 και τη 3. Τα φάρμακα εξαιρούνται όμως. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να περάσει από μια αναθεώρηση του κανονισμού για να προσθεθούν και τα φάρμακα που περιέχουν εφεδρίνη και ψευδοεφεδρίνη που είναι οι βασικές πρόδρομες ουσίες των μετααμφεμινών και θεωρούνται σαν ουσίες επικίνδυνες. Οι ουσίες αυτές όμως είναι εύκολο να αφαιρεθούν από τα φάρμακα μέσα στα οποία κυκλοφορούν. Τα φάρμακα αυτά είναι πάρα πολύ κοινά. Χρησιμοποιούνται εναντίον των αλλεργιών, εναντίον της γρήπης, του συναχιού κτλ. Στόχος λοιπόν της αναθεώρησης είναι τα φάρμακα αυτά να μπουν στο πεδίο κανονισμού και να δώσουν στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών την δυνατότητα αντιμετώπισης της καταχρηστικής τους μεταχείρισης. Είναι σωστή η στόχη αυτή της αλλαγή. Διαρωτώ με όμως για το πόσο είναι, ε, θα έλεγα, έγκριτο το πεδίο εφαρμογή που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εξαιρούνται τα φάρμακα. Κανένα φάρμακο δεν μπορεί να προσθεθεί στο παράρτημα σαν ταξινομημένη ουσία στις τρεις κατηγορίες. Γι' αυτό δημιουργεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα σύστημα sui generis που εφαρμόζεται ειδικά στα φάρμακα με εφεδρίνη και ψευδοεφεδρίνη. Αυτό είναι κάτι που δημιουργεί θέματα για μένα. ένα ειδικό καθεστώς θα δημιουργήσει προβλήματα και στο ευανάγνωστο του κειμένου. Οι ουσίες μπορεί να προσαρμοστούν. Οι κατάλογοι αυτοί έτσι και αλλιώς τροποποιούνται με ε, εξουσιοδότηση πράξης, κάτι το οποίο επιτρέπει μια κάποια ευελιξία. Αλλά αν αφαιρεθούν τα φάρμακα και από τα παραρτήματα, είναι κάτι που επιβάλλει τη συναπόφαση για την παραμικρή τροποποίηση. Αν σαν παράδειγμα συνειδητοποιήσουμε ότι το σύστημα sui το οποίο δημιουργήθηκε για την εφεδρίνη και την ψευδεφεδρίνη, είναι λιγότερο αποτελεσματικό από τα προηγουμένως ισχύοντα. Αυτό θέλουμε. Και τι θα συμβεί αν οι έμποροι ναρκωτικών βρουν κι άλλο ένα φάρμακο από το οποίο μπορούν να βγάλουν μια πρόδρομο ουσία γρήγορα και εκεί θα πρέπει να περνάμε από τη συναπόφαση που είναι μια διαδικασία η οποία είναι γραφειοκρατική και ε, μακρόπρονη. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα. Κατανοώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει ένα ειδικό καθεστώς για τα φάρμακα. Αλλά δεν θα μπορούσαμε να βρούμε ένα διαφορετικό σύστημα εκτός από το ειδικό καθεστώς για ένα φάρμακο ένα σύστημα το οποίο να επιτρέψει μεγαλύτερη δυνατότητα αντίδρασης. Γιατί δεν μπορεί να περιμένουμε δύο χρόνια για να προσαρμοστούμε όπως αυτό θα ίσχυε στην περίπτωση της συναπόφασης. Αυτό δεν είναι σοβαρό. Δεν θα έχουμε υιοθετήσει το έγγραφο και οι έμποροι ναρκωτικών θα βρούνε μια διαφορετική λύση. Μήπως θα μπορούσαμε λοιπόν να βρούμε μια τέταρτη κατηγορία στα παραρτήματα. Αν τα φάρμακα ανήκουν σε ένα ειδικό καθεστώς, την οδηγία 2001-83, αυτό το κάνουν ε, λόγω των επιπτώσεών του στην υγεία. Και η διάδοση των ναρκωτικών επίσης επηρεάζει την υγεία πολλών πολιτών. Είμαι υπέρ λοιπόν μιας άλλης λύσης, η οποία θα επιτρέψει μεγαλύτερη και γρηγορότερη δυνατότητα αντίδρασης αν βρεθούν στις αγορές και διαφορετικές φαρμακευτικές ουσίες από την εφεδρίνη και ψευδοεφεδρίνη. Μία τεχνική ερώτηση τώρα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη σύνδεση των άρθρων 11 και 12 όπως έχουν τροπολογηθεί. Το 11 στην παράγραφο 1 λέγει ότι οι εξαγωγές ουσιών κατηγορίας 3 ορισμένες χώρες θα πρέπει να συνοδεύονται από μία συγκεκριμένη ανακοίνωση ε, προς εξαγωγή. Το άρθρο 12, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 3, λέγει ότι οι ουσίες που ταξινομούνται στην κατηγορία 3 υπόκεινται σε μία εκ των προτέρων αδειοδότηση για εξαγωγή, εφόσον έχει υπάρξει ειδική διακίνωση ή εφόσον ε, εξάγονται σε χώρες οι οποίες περιλαμβάνονται στο, παράδειγμα, στο παράρτημα. Οι ουσίες αυτές πράγματι συνοδεύονται από τέτοιου είδους ε, έγγραφα για τις εξαγωγές, ακριβώς γιατί εξάγονται στις συγκεκριμένες χώρες. Γιατί λοιπόν να υπάρχει αυτή η επικάλυψη ανάμεσα στα δύο άρθρα. Τώρα το δεύτερο σημείο, η επιτροπολογία, η οποία είναι κάτι το πολύ πιο απλό θα έλεγα, μη σας ανησυχεί. Όπως είπα πριν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εποφελείται από την αναθεώρηση αυτή για να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της νέας συνθήκης για την επιτροπολογία. Γενικά η μεταφορά εδώ αρμοδιοτήτων τεκμηριώνεται στις περισσότερες από τις περιπτώσεις. Πιστεύω όμως ότι στο 30 α μικρό η Επιτροπή δεν διευκρινίζει τι θέλει. Λέει ότι μπορεί να υιοθετήσει κατεξουσιοδότηση πράξης για να προσαρμοστεί στις νέες τάσεις σε σχέση με την καταχρηστική μεταχείριση των ουσιών αυτών. Στο 33 επίσης λέγεται ότι η δυνατότητα αυτού του χαρακτηρισμού μπορεί να είναι αορίστου διαρκείας, κάτι το οποίο βρίσκω ότι είναι υπερβολικό. Θα κάνω μια διαφορετική λοιπόν εγώ πρόταση για τη διάρκεια της αδειοδότησης κατ' εξαίρεση με δυνατότητα παράτασης άμα τη λήξη της. Εγώ θα ήθελα λοιπόν να επιλέξουμε την διαβούλευση η οποία επιτρέπει πιο ταχεία και αποτελεσματική αντίδραση με πιο αποτελεσματική ε, ταυτόχρονα καταπολέμηση των ναρκωτικών ουσιών. Είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστούμε κύριε Σιγητά. Ελπίζω η Κομισιόν να έχει σημειώσει τις περιστατωμένες σκέψεις, επιφυλάξεις και αντιδράσεις του εισηγητή. Πάμε τώρα στους σκιώδεις. Μόνο η Φρανσίσκα Κέλλερα από Πράσινους είναι εδώ, οπότε της δίνω το λόγιο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και τον εισηγητή. Έχω και εγώ κάποιες ερωτήσεις και κάποιες πολύ σχετικά με αυτή την πρόταση προς την Κομισιόν αναφέρατε ότι περίπου 600 κιλά αυτών των ουσιών ε, δεσμεύτηκαν από τις αρχές το 2009. Θα ήθελα όμως να γνωρίζω πόσα κιλά ή τόνοι ε, είναι το συνολικό εμπόριο, δηλαδή το προβληματικό κομμάτι. Αυτό είναι σημαντικό για να κατανοήσουμε το μέγεθος του προβλήματος που έχουμε εδώ. Επιπλέον, αναφέρατε ότι θέλετε να είναι πιο δύσκολο, πιο ακριβό και πιο επικίνδυνο για τους εγκληματίες ε, να κατασκευάζουν ε, ναρκωτικά. Όμως ε, αυτή η δαπάνη πόσο θα επιβαρύνει τις εταιρείε που θα χρησιμοποιούν νόμιμα αυτές τις ουσίες για τα φάρμακά τους. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω κάποια πράγματα γι' αυτό επιπλέον. Επίσης είπατε ότι δεν θέλετε να έχουμε εμπόδια σε επίπεδο ε, νόμιμου εμπορίου, πώς θα διασφαλίσετε ότι αυτό θα γίνει και πώς θα αξιολογήσετε τις επιπτώσεις της πρότασης ε, στο νόμιμο εμπόριο. Θα υπάρχουν κάποιες ε, καθυστερήσεις στο νόμιμο εμπόριο. Για παράδειγμα, στο εμπόριο φαρμάκων. Θα υπάρχει κάποια καταχώρηση, κάποιος έλεγχος κατά την εξαγωγή πόσο θα καθυστερήσει δηλαδή το νόμιμο εμπόριο φαρμάκων όπου οι καθυστερήσεις αποτελούν πρόβλημα. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου. Έφτασε η Σκιώδης ε, Χωσέφ Ανδρέας από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά ήρθα από μία άλλη συνεδρίαση σε μια άλλη επιτροπή. Η τροποποίηση του κανονισμού για τον έλεγχο των ουσιών σε επίπεδο τελωνιακό ορισμένων φαρμάκων που περιλαμβάνουν αυτές τις πρόδρομες ουσίες είναι ένα θέμα. Υπάρχει μια κάποια μεγάλη ανησυχία για την εμπορία των ναρκωτικών ουσιών Η συνθήκη της Λισαβόνας δίνει αρμοδιότητα τέτοια και στο Κοινοβούλιο. Και έχουν υπάρξει αρκετές εκθέσεις και έχουν προηγηθεί πολλές συζητήσεις ε, για τις ε, κατηγοριοποιήσεις ε, και τα διάφορα είδη ναρκωτικών. Η ηρωίνη, κοκαίνη, συνθετικά ναρκωτικά κτλ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για φάρμακα τα οποία περιλαμβάνουν ουσίες όπως η εφεδρίνη και η ψευδοεφεδρίνη που μέσω τεχνικής επεξεργασίας σχετικά απλής και εύκολης ε, μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή μεταμφεταμίνης, η οποία είναι πάρα πολύ ε, ζητούμενη ναρκωτική ουσία και προκαλεί επιπτώσεις άμεσα. Κανονικά θα πρέπει οι χώρες να ελέγχουν τα, τις ουσίες αυτές, όχι όμως σε τελωνιακό επίπεδο. Ε, σε αυτό το επίπεδο δεν είναι δυνατό να ελέγχονται οι αποστολές των φαρμάκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των φαρμάκων όταν εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να έχουν κάποια μέσα στη διάθεσή τους οι τελωνιακές αρχές, ε, μέσα που να βασίζονται πρώτον στο θέμα της ε, των συνοδευτικών εγγράφων όταν υπάρχει μια σημαντική αποστολή τέτοιων φαρμάκων ή να υπάρχει ένας κατάλογος ε, στον οποίο να εγγράφονται υποχρεωτικά τα φάρμακα αυτά αλλά είναι σαφές ότι σε αυτή τη φάση τα τελωνία δεν είναι σε θέση να κάνουν αυτούς λοιπόν αυτές τις δυνατότητες, πρέπει να έχουν τις δυνατότητες αυτές, πρέπει να διορθωθεί ένα λάθος το οποίο υπάρχει και έχω την εντύπωση ότι ακριβώς και σε συνεργασία μεταξύ των πολιτικών ομάδων μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα αποτελεσματικό θα έλεγα έγγραφο έτσι ώστε τα φάρμακα αυτά και να ελέγχονται καλύτερα και να βελτιωθεί φυσικά και η δημόσια υγεία. Πριν δώσω το λόγο στην Κομισιόν, να ακούσουμε λίγο και τον εισηγητή σχετικά με την επιτροπολογία. Δεν ξέρω εξ αρχής γιατί η Κομισιόν υποχωρεί στη θέση του Συμβουλίου και αρχίζει ε, προτείνοντας μια τέτοια διαδικασία εξέτασης. Όντως ε, υπάρχει ο κανόνας στη συνθήκη όταν ε, υπάρχει επιτροπολογία να υπάρχει μια συγκεκριμένη μητρά εξέτασης. Όμως υπάρχουν και εξαιρέσεις. Νομίζω ότι είναι τόσο σημαντικό το θέμα που θα έπρεπε να υπάρχει βέτο. Γιατί η Κομισιόν να μην παλεύει πιο πολύ για την αυτονομία των κρατών μελών όταν μιλάμε για ευρωπαϊκή νομοθεσία και εκ μέρους της Κομισιόν το Κοινοβούλιο να έρχεται και να υπερασπίζεται την αυτονομία της Κομισιόν. Πραγματικά με εκπλήσει. Δεν θα πρέπει να υπάρχει βέτο. Η Κομισιόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Καλημέρα, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Προύστ για την δουλειά που έχει κάνει πάνω σε αυτή την πρόταση της Κομισιόν. Χαίρομαι που υπάρχει συνολική υποστήριξη στους στόχους που προσπαθούμε να πετύχουμε με αυτή την πρόταση. Πραγματικά δημονούμε για μια ενδιαφέρουσα συζήτηση σχετικά με το πώς θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε αυτό το κείμενο, το οποίο ε, δεν αντιμετωπίζει μάλλον όλα τα ανοιχτά θέματα. Για το πρώτο σημείο, την εξαίρεση φαρμάκων από το πεδίο του κανονισμού, αυτή είναι μια κατάσταση που έχουμε κληρονομήσει από τον κανονισμό. Όπως ξέρετε, το εμπόριο των φαρμάκων ε, ρυθμίζεται από μια οδηγία η οποία πρόσφατα τροποποιήθηκε και δεν θεωρήσαμε ότι υπήρχε ανάγκη να καλυφθούν αυτά τα προϊόντα και με αυτόν τον κανονισμό αν δεν υπάρχουν πρόδρομες ουσίες σε αυτά. Στα περισσότερα φάρμακα, σε, όλες, σε όλα σχεδόν που καλύπτονται από την πρόταση, δεν υπάρχουν πρόδρομες ουσίες που εύκολα εκχυλίζονται από τους ε, ε, εμπόρους ναρκωτικών. Και γι' αυτό το λόγο προτείναμε συγκεκριμένη διάταξη για αυτά τα φάρμακα που περιέχουν εφεδρίνη και ψευδοεφεδρίνη. Τα γνωρίζετε αυτά. Όταν έχουμε βήχα τα παίρνουμε. Είναι σε σκόνη πολύ συχνά. Μπορείτε να δείτε συνταγές στο ίντερνετ για την εκχύληση της ψευδοεφεδρίνης από αυτά τα φάρμακα. Έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή στην αγορά υπάρχουν ε, φάρμακα τα οποία μπορούν ε, εύκολα να μας δώσουν πρόδρομες ουσίες και να παραμείνει σταθερή ουσία. Είμαστε λοιπόν στην εξής κατάσταση. Θέλουμε να βρούμε μια συγκεκριμένη διάταξη για τα συγκεκριμένα αυτά φάρμακα. Ο στόχος επίσης είναι να μην ε, εμποδίσουμε το νόμιμο εμπόριο σε φάρμακα και αυτή θα είναι και η πιο λογική προσέγγιση προς αυτή την κατεύθυνση. Η εξαίρεση ε, των φαρμάκων από τον ορισμό είναι σημαντικό κομμάτι της πρότασης, γιατί καλύπτει όλο το πεδίο, γι' αυτό δεν ζητήσαμε εξουσιοδότηση ε, για την Κομισιόν να βάλει επιπλέον ε, φάρμακα στο παράρτημα. Για τη σχέση μεταξύ του άρθρου 11 και 12, όντως ξαναδιαβάσαμε τις διατάξεις και η ιδέα είναι ότι ε, υπάρχουν ε, κάποιες ουσίες ε, που χρειάζονται μια τέτοια ένα έντυπο κοινοποίησης εξαγωγής και όταν υπάρχει ένα τέτοιο έντυπο, καλό θα είναι να βελτιώνεται η διατύπωση για να είναι ξεκάθαρο ξεκάθαρη. Για το άρθρο 13α εξουσιοδότηση στην Κομισιόν για να μπορέσει να τροποποιήσει το παράρτημα ώστε να αντιδρά σε νέες τάσεις. Εδώ ε, η πρόθεση ήταν όταν βλέπουμε ένα νέο προϊόν το οποίο δεν έχει ξαναχρησιμοποιηθεί στο παρελθόν να χρησιμοποιείται για να παρακάπτονται οι έλεγχοι για τις πρόδρομες ουσίες, να μπαίνει στον κατάλογο αμέσως η ουσία. Αυτός ήταν ε, ο στόχος, ε, η αντιμετώπιση νέων τάσεων στο παράνομο εμπόριο. Θέλαμε να είναι λίγο γενικό για να μπορεί να καλύπτει τις τάσεις που δεν μπορούμε από τώρα να περιγράψουμε. Αυτό που είπαμε όμως ε, επίσης είναι ε, ότι είναι για ουσίες από τις οποίες εύκολα ε, μπορεί κανείς να λάβει τις πρόδρομες ουσίες. Αυτό διασφαλίζεται με την πρόταση. Όπως είπε ο κύριος Προύστ, είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της πρότασης και νομίζω ότι όλες οι αρχές στα κράτη-μέλη πραγματικά προσμένουν την δυνατότητα της Κομισιόν να αντιδρά πιο γρήγορα σε νέες παράνομες ουσίες. Τώρα, να απαντήσω στις ερωτήσεις για το εμπόριο. Για τον όγκο του εμπορίου. Σήμερα δεν έχουμε στατιστικές για τον όγκο αυτών των ουσιών που υπάρχουν στο εμπόριο οι στατιστικέ του διεθνού εμπορίου δεν έχουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, το, για το ε, διεθνές εμπόριο υπάρχει ένα κοινό και εναρμονισμένο σύστημα και ονοματολογία. Δεν υπάρχει όμως συγκεκριμένος δοσμολογικός κώδικας ε, για την κατάταξη ε, φαρμάκων με εφεδρίνη και ψευδοεφεδρίνη, καλύπτονται από έναν γενικότερο κωδικό. Γι' αυτό το λόγο στο μεταξύ προτείναμε τη δημιουργία ενός συγκεκριμένου κωδικού για αυτές τις ουσίες στην συνδυασμένη ονοματολογία και ζητήσαμε τον Παγκόσμιο Οργανισμό ε, Δασμών να τις ε, συμπεριλάβει στο ε, τελωνίων μάλλον να το συμπεριλάβει στο κατάλογό του και γι' αυτό θα μπορέσουμε να έχουμε και καλύτερες στατιστικές για αυτό το θέμα. Τώρα, όσον αφορά στις επιπτώσεις της πρότασης ε, ε, στις ε, εταιρείε, πρόκειται για αυτό το έντυπο κοινοποίηση της εξαγωγής, έχουμε ειδοποιήσει τον σύνδεσμο της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας Φαρμάκων και έχουμε κάνει μια διαβούλευση θεωρούν ότι θα είναι ελάχιστες οι επιπτώσεις ε, στο εμπόριο και στις συναλλαγές, γιατί αυτή η κοινοποίηση πριν από την εξαγωγή είναι ουσιαστικά οι πληροφορίες που θα δίνουν στην χώρα εξαγωγή οι αρχές ε, της χώρας ε, που εξάγει. Υπάρχει ήδη λοιπόν αυτή η υποχρέωση από την πλευρά της εταιρείας. Δίνει λοιπόν στο τελωνία αυτή την ε, δήλωση για την εξαγωγή. Μετά ε, αποστέλλεται η κοινοποίηση στη χώρα ε, που θα πάει η εξαγωγή και μέσα σε 15 μέρες η χώρα που θα εισάγει το φάρμακο πρέπει να απαντήσει σχετικά με το κατά πόσο είναι εντάξει διαδικασία. Οπότε ο κανονικός χρόνος για την εξαγωγή φαρμάκων ε, είναι ε, λίγο πολύ ο ίδιος. Δεν νομίζουν ότι θα έχουν λοιπόν οι εταιρείε επιπλέον επιβάρυνση στις συναλλαγές τους. Επιπλέον, η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη θα επαγρυπνούν έτσι ώστε το σύστημα να μην ε, δημιουργεί καθυστερήσεις στο νόμο εμπόριο. όχι μόνο για τις ε, κοινοποίησεις αυτές πριν από την ε, ε, εισαγωγή, εξαγωγή, αλλά και για τους ελέγχους στα τελωνία. Απάντησα νομίζω τις περισσότερες ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Δεν απαντήσατε στη δική μου ερώτηση. Κουφ ήταν μια επανάληψη μια ερώτηση που έθεσε ο ίδιος ο εισηγητής. Γιατί η επιλογή ε, η Επιτροπή επέλεξε αυτή τη διαδικασία εξέτασης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν είχα σκοπό να μην απαντήσω. Προτίσαμε τη διαδικασία εξέτασης ε, με βάση τους γενικούς κανόνες ε, που ακολουθούνται σε θέματα εμπορικής πολιτικής. Να πω όμως επίσης ότι όλη η νομοθετική και επιχειρησιακή δουλειά που κάνουμε σήμερα είναι ε, μία συνεργασία μεταξύ της βιομηχανίας, των αρχών των κρατών μελών και της Κομισιόν. Γι' αυτό το λόγο, όταν ε, προτείνουμε την προσθήκη μιας ουσίας σε παράρτημα, είναι πολύ σημαντικό για εμάς να έχουμε πληροφορίες από τους εμπειρογνώμενους των κρατών μελών. Γι' αυτό ξεκινήσαμε με αυτή τη διαδικασία, αλλά φυσικά είμαστε ανοιχτοί προς εναλλακτικέ. Δεν χρειάζεστε μόνο πληροφορίες από αυτούς, αλλά και τη συμφωνία τους. Τη συμφωνία τους. Ο εισηγητής έχει το λόγο. Μία διευκρίνηση θα ήθελα να κάνω για να απαντήσω στις ερωτήσεις. Άκουσα τα λόγια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα συνεργαστούμε βέβαια, θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας. Δεν υπάρχει ιδανική λύση ως προς την ταξινόμηση. Το μη βέλτιστον. Αυτή τη θέση να υιοθετήσουμε και να φτάσουμε σε μια νέα ταξινόμηση. Γνωρίζουμε ποια είναι η κατάσταση σήμερα με τα φάρμακα αυτά, με αυτές τις φαρμακευτικές ουσίες, αλλά δεν ξέρουμε ποιο είναι το αποτέλεσμα ε, ποιο έχει σχέση ε, π.χ. το ακετατικό οξύ με την βιομηχανία του ξυδιού. Είναι δύσκολο. Αυτό είναι το η δυσκολία της έκθεσης. Δηλαδή, να μην υψώσουμε εμπόδια στην εμπορική δραστηριότητα, αλλά απ' την άλλη να είμαστε αποτελεσματικοί ως προς τις πρόδρομες ουσίες. Βασικό μας μέλημα πρέπει να είναι να μην υπάρξουν δυσκολίες σε υπερ... διότι όταν αποφασίζουμε κάτι με συναπόφαση αυτό παίρνει πάρα πολύ χρόνο και είναι δύσκολο να έχει αναδρομική ισχύ και ως προς την επιτροπολογία αυτή η διαδικασία διαβούλευσης είναι, ε, δεν είναι τόσο κατάλληλη όσο η διαδικασία εξέτασης. Άρα η έκθεση αυτό το στόχο έχει, να μην σβήσει η εμπορική δραστηριότητα σε αυτούς τους κλάδους της οικονομίας, αλλά από την άλλη να μπορούμε να ασκούμε, να κάνουμε τους ελέγχους μας, ώστε να έχει επιτυχία ο αγώνας μας κατά των ναρκωτικών ουσιών. Ε, αυτή είναι η δυσκολία του. Πώς θα συγκεράσουμε τα δύο αυτά πράγματα. Ευχαριστώ πολύ, ο Πρόεδρος. Και εγώ σας ευχαριστώ. Θα εξετάσουμε το σχέδιο της έκθεσης την επόμενη φορά που θα συνεδριάσουμε ως Επιτροπή, 20 και 21 Φεβρουαρίου. Επομένως, ο συνάδελφος Φρανκ Προύστ θα μας υποβάλει σε εύθετο χρόνο το σχέδιο της έκθεσης για να το εξετάσουμε τότε. Ε, να κάνουμε ενδεχομένω ένα διάλειμμα θα έχουμε συνεδρίαση των συντονιστών. Όσοι δεν έχετε δικαίωμα να ε, παραστείτε στην αίθουσα, παρακαλώ να αποχωρήσετε. Μπορείτε να φύγετε, είστε ελεύθεροι. Θα συνεχίσουμε την συνεδρίαση σήμερα το απόγευμα ως Επιτροπή. Οι συντονιστές συμφώνησαν να ξεκινήσουν νωρίτερα στις 11 και 4. Επομένως, σε 15 λεπτά ξεκινάμε πάλι.